Καλημέρα σας. Μας δώσαν τη μεγαλύτερη αίθουσα επιτροπή σήμερα. Τι τιμή. Συγγνώμη που υπάρχει λίγη... Υπάρχει... Ακούμε λίγη ηχό στην αίθουσα. Θα θέλω να ευχαριστήσω και όσους μας ακούν από το διαδίκτυο. Θα έχουμε μία ε, σειρά συνεδριάσεων και στο τέλος του μήνα μετά από την επόμενη εβδομάδα, μετά από την Ολομέλη. Θα ήθελα να αλλάξουμε κάτι στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί λόγω της διαθεσιμότητας των ε, εισηγητών για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και για τα επενδυτικά προϊόντα να τα πάμε στο τέλος, 11.30 ώρα και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την προστασία των επιχειρήσεων κατά των παραπλανητικών πρακτικών marketing. Αυτά. Επειδή θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο σήμερα με αυτά, να τα πάμε στην θέση των, άλλων, των προηγούμενων θεμάτων. Οπότε Αυτά ήθελα να σας πω για τις αλλαγές της ημερήσιας διάταξης. Πριν περάσουμε στην ουσία της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να σας πω ότι πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στην Κροατία πάρα πολύ καλή συνάντηση. Συναντήσαμε τον κύριο Νίμιτσα που είναι ο αντιπρόεδρος της ε, κυβέρνησης της Κροατίας και άλλους υπουργούς και είχαμε, μια, είχαμε πολύ διεξοδικές και περιεκτικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις καταναλωτών. Επίσης καταφέραμε να πάμε όχι μόνο στο Ζάγκρεπ αλλά και στο Σπλίτ που είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με προσώπους τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι συνεδριάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ε, συνάδελφο που μας βοήθησε τόσο πολύ Μάτιτς, τη συνάδελφο Μάτιτς που μας βοήθησε τόσο πολύ να τα οργανώσουμε όλα αυτά και να έχουμε το μέγιστο αριθμό συναντήσεων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και επίσης φύγαμε πολύ αργά από το Ζάγκρεπ για να πάμε στο Σπλίτ και φτάσαμε όλοι, δεν έμεινε κανείς πίσω, τα καταφέραμε. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως, ε, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό μετά. η... τα πρακτικά της 20 ε, και 21 Φεβρουαρίου και της 4 Μαρτίου 2013 θα θεωρηθούν εγκεκριμένα μέχρι το τέλος συνεδρίασης αν δεν υπάρξουν ε, αντιρρήσεις. Από εδώ και στο εξή, σε κάθε συνεδρίαση θα γίνεται μια ενημέρωση και για του ευρωβουλευτέ αλλά και για το κοινό για σημαντικέ διαπραγματεύσει, που συμμετέχει η Επιτροπή μα ε, για συμφωνίε σε πρώτη ανάγνωση Είχαμε δύο συναντήσεις τριμερή, σε τριμερή διάλογο αυτή τη βδομάδα και θα έχουμε και άλλες ε, την επόμενη βδομάδα. Όλοι οι συγητές λοιπόν είναι πάρα πολύ απασχολημένοι, όπως και εγώ και το προσωπικό της Επιτροπής. Το χρονοδιάγραμμά μου λοιπόν είναι πολύ πιεσμένο. Κάνουμε όμως ε, πολύ σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον Φιλίπ Ζουβά να μας πει ορισμένα πράγματα για το δικό του θέμα και μετά θα περάσουμε στην κυρία Γκέπχαρτ ε, για, εκ μέρους κυρίου Ταραμπέλα για τις δημόσιες προμήθειες. Μετά επίσης θα μιλήσουμε για τις επαγγελματικές δεξιότητες. Έχουμε το πακέτο ευθυγράμμισης της κυρίας Ροϊτόβα και τον τελωνιακό κώδικα, τον οποίο θα τον παρουσιάσω εγώ εκ μέρου του συναδέλφου που λείπει. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ας ακούσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα από τους συζητητές. Κύριε Ζουβάν, σας καλώ να, μας, να αρχίσετε την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για τις ε, για τις ε, συμβάσεις παραχωρήσεων. Έγινε ε, μία συνεδρίαση χθε, θα γίνει και σήμερα το απόγευμα. Έγιναν αναλύσεις ε, του κειμένου παράγραφο προς παράγραφο. Εκτός από τα 11, 15 και 11α άρθρα, μέχρι το άρθρο 40, γιατί υπήρχαν κάποια κοινά σημεία με τις δημόσιες προμήθειες και προτάθηκαν συμβιβασμοί στο Συμβούλιο χθε. έγινε η δεύτερη επίσημη συνάντηση τριμερούς διαλόγου η πρώτη ήταν ε, παρατήρηση ε, συνάντηση, οι ΜΕΝ και οι ΔΕ ανέφεραν τις θέσεις τους και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον ευγενικά. Ε, μιλούσαμε για τα διάφορα κείμενα που είχαμε μπροστά μας, όμως ε, εχθές τα πράγματα πήγαν πολύ καλά εχθές ε, στην εξέλιξη της ε, συνάντησης γιατί το, το Συμβούλιο δέχθηκε κάποιους από τους συμβιβασμούς. Οι συμβιβασμοί δεν είναι επίσημοι ακόμη, αλλά η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε ικανοποιητικό κείμενο και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Κάποια συγκεκριμένα ζητήματα βέβαια χρήζουν συζήτηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών, ε, ο οικονομικός κίνδυνος για παράδειγμα πώς ορίζουμε αυτόν τον κίνδυνο ικανοποιητικά. Το κατόφλι επίσης μπορούμε να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν τα 5 έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ και το ζήτημα του αντικτύπου των διεθνών ε, συμβάσεων. Είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των σκιωδών πριν από την συνάντηση με το Συμβούλιο. Καλά πάνε πάντω τα πράγματα και μπορούμε να ελπίζουμε ότι κατά τις επόμενες ημέρες ε, θα ε, υπάρξουν και επίσημες συμφωνίες. 25 Απριλίου είναι ο επόμενος τριμερής διάλογος και θα συζητηθούν μεταξύ άλλων ε, οι τομεακές εξαιρέσεις άρθρο 8, κοινωνικές υπηρεσίες άρθρο 17 και η διακυβέρνηση άρθρο 43. 11α είναι ένα σημαντικό άρθρο από πολιτική απόψεως γιατί θα θυμάστε ότι μας είχε δοθεί εντολή να διαπραγματευτούμε με παρέμβαση ε, του Επιτρόπου για τη βάση ε, των ζητημάτων ε, υδάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη Πρέπει όμω να μιλήσουμε πρώτα για το 11, γιατί το 11α αποτελεί ουσιαστικά μία εξαίρεση στο 11 και θα ήταν περίεργο να το συζητήσουμε πρώτο. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να εξευρεθούν λύσει. Το 11 πρέπει να συζητηθεί, το 15 επίση, σε έναν τριμερή ε, διάλογο με, ε, τους, ε, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει να μιλήσουμε για το 11 και το 15 με τους συναδέλφους για τις δημόσιες προμήθειες και μετά να μιλήσουμε για το θέμα 11α που είναι οι εξαιρέσεις που γνωρίζετε μετά από αυτό τον τριμερή διάλογο. Το λέω αυτό για λόγους ημερήσιας διάταξης, κάπως πρέπει να τα συμβιβάσουμε, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα πηγαίνουν μάλλον καλά. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας, ενθαρρυντική η αναφορά αυτή και νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς υπάρχουν κάποια κοινά σημεία που θα έχουμε κοινό τριμερή διάλογο μεταξύ κυρίων Τεραμπέλα και Ζουβάν. Θα έχουμε κάποιες κοινέ ρήτρε λοιπόν. Να προχωρήσουμε στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, κυρία Γκέπαρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προχωρήσω μιλώντας γαλλικά, γιατί ο κύριος Ταραμπέλα μου έδωσε τις σημειώσεις του στα γαλλικά και είναι πιο εύκολο. Και συμφωνεί ο κύριος Ταραμπέλα με τον κύριο Ζιβέν για να συζητηθούν τα άρθρα 15 και 11 και τα υπόλοιπα ε, σε μια κοινή συνεδρίαση, γιατί πρέπει να δράσουν έτσι έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση στα δύο θέματα αυτά γιατί βρίσκονται πολύ κατά το ένα στο άλλο. Και τώρα φτάνω στον τριμερή διάλογο για τις δημοσίες συμβάσεις. Στις 26 Μαρτίου έλαβε χώρα τελευταίος τριμερής διάλογος, η συζήτηση στην ημερησία διάταξη, ίσως αντικείμενο, τα κλάστερ 5 και 2, σε δύο άρθρα, στο άρθρο 44, σε ό,τι αφορά την οικονομία και το 15.2, σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό σεβασμό κοινωνικών κριτηρίων και σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις δεν είχαμε συζήτηση βάθος, μόνο ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Θα μπούμε περισσότερο στις ε, ε, λεπτομέρειες για τις παραγράφους στο Plan Explain ε, και αυτό έχει να κάνει με το να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στη συζήτηση του άρθρου 56.3 σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική δυνατότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την πρόσβαση σε μια σύμβαση, συμφώνησε το Κοινοβούλιο να μειωθεί η αξία από τρει σε δύο φορές ε, στην αξία της σύμβασης ε, και να λάβει υπόψη την εκφερεγγιότητα της το Συμβούλιο όμως ε, στο θέμα αυτό δεν έδειξε να υποχωρήσει το άρθρο 15.2 η συζήτηση ήταν ουσιαστική. Το Κοινοβούλιο είπε ότι το άρθρο αποτελεί κόκκινη γραμμή η Κομισιόν ε, είπε ότι δέχεται τις γενικές αρχές, ενώ το Συμβούλιο παραμένει ιδιαίτερα διστακτικό. Στο άρθρο 54.2, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να υπάρχει τροποποίηση των φάσεων επιλογής, ε, το Κοινοβούλιο ε, ζήτησε να υπάρχουν αυστηρά μέτρα για την εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού, καθώς και την ομοιόμορφη μεταφορά

στο εσωτερικό δίκαιο όλων των χωρών σε ό,τι αφορά τις ε, ε, ιδιαίτερα χαμηλές προσφορές ε, το Κοινοβούλιο έχει την υποστήριξη της Ομισιόν κατά του Συμβουλίου για να υπάρχει υποχρέωση από την του αρχή για να ζητήσει την αιτιολογία. Αν το Κοινοβούλιο άδειασε το περιεχόμενο του άρθρου, το Κοινοβούλιο παραμένει πεπισμένο για την αναγκαιότητα καταπολέμησης ε, του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμητου ανταγωνισμού Δίνοντα στην αναθέτηση αρχή τα απαραίτητα εργαλεία. Για το άρθρο 55.1, κριτήρια αποκλεισμού, είχαμε μία συμφωνία για μία αλλαγή στην διατύπωση αλλά υπάρχει αντίρρηση του Κοινοβουλίου στις παρεκκλήσεις ε, που γίνονται εξ ονόματος του Γενικού Συμφέροντος ε, γιατί είναι αόριστες και αδιαφανείς. Όλοι οι συγητές δήλωσαν διαθεσιμότητα να κάνουν εξαιρέσεις για το κριτήριο αποκλεισμού. Μόνο η διατύπωση αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως πρέπει να χάρη στη η συζήτηση του άρθρου 66 ως ε, το μόνο κριτήριο ανάθεσης ε, ε, εκεί το Κοινοβούλιο έχει μια συγκεκριμένη θέση, αλλά υπάρχει αντίθεση από τα άλλα όργανα. Στο άρθρο 67 ε, το, πρέπει να ξανασυζητηθεί το άρθρο αυτό σε σχέση με το κόστος, αλλά θεωρούμε ότι το κείμενο του Συμβουλίου αποτελεί μια καλή βάση αφετηρία. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προσεγγίσει, αλλά ε, με την ε, εξαίρεση του κειμένου για τους εξωτερικούς παράγοντες. αυτά συζητήσει κάνουμε με τον κύριο Τεραμπέλα για του τομεί αυτού. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση πηγαίνει καλά και όπω είπα στην αρχή και το επαναλαμβάνω, ο κύριο Τεραμπέλα συμφωνεί για να γίνει μια κοινή συζήτηση για τα άρθρα 15 και 11 για τις συμβάσεις παραχώρησης. Από την αρχή λέει το Κοινοβούλιο ότι είναι μια κοινή δεσμή μέτρων και θα προτιμούσε να μην ε, διαιρέσει τα γιατί πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των κειμένων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τώρα, επί τη ευκαιρία, θα δεχτώ ερωτήσεις από εσάς όταν τελειώσουμε με όλες τις εκθέσεις. Και τότε θα, μπορείς, θα μπορείτε να ρωτήσετε τους εισηγητές. Τώρα, ο κ. Φανιού δεν είναι εδώ. Και νομίζω ότι από την τελευταία έκθεση δεν είχαμε τριμερή διάλογο. Όταν έρθει λοιπόν θα την καλέσω να λάβει το λόγο. Να πω όμως ότι ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 24 Απριλίου. Αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε μόνο έναν τριμερή διάλογο στις 20 Μαρτίου. Χρειαζόμαστε και άλλον. Όπως και με όλους τους φακέλου υπάρχει πολύ μεγάλη δουλειά πρέπει να γίνει, τεχνική φύση. Και πιστεύω πως ε, δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος πόσο πολύ και πόσο τεχνική είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Το Συμβούλιο κάνει πάρα πολλές τεχνικές αλλαγές στα κείμενα και εμείς φυσικά πρέπει να τις εξετάσουμε λεπτομερώς. Και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, έτσι ώστε να γίνει σωστή δουλειά. Προχωράμε τώρα. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το πρώτο πακέτο στο Συμβούλιο Αγκρή συζήτησε ορισμένα άρθρα. Και τώρα η συνάδελφος θα μας ενημερώσει για τις συζητήσεις για το πακέτο ευθυγράμμισης. Τώρα, για τα, για τα σκάφη αναψυχής, μπορώ να σας πω ότι αρκετές από τις τροπολογίες μας εγκρίθηκαν και πιστεύω πως ε, στην επόμενη συνεδρίαση στο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο θα καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, πολλές τροπολογίες μας έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση του Συμβουλίου μετά από τις αρκετά τεχνικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα με εμπειρογνώμονες. Τώρα, όσον αφορά τον τελωνιακό κώδικα. Βρέθηκα σε συνεδρίαση με την κυρία Λεγκρίπ, η οποία δυστυχώς δεν είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της. Έγινε λοιπόν ο τριμερής ε, διάλογος την Τρίτη το πρωί. Και αυτό το πακέτο είχε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες τώρα έγιναν επισήμως δεκτές. Έγινε μεγάλη πρόοδος στα πολιτικά στοιχεία του φακέλου, όμως ακόμα υποβάλλουμε συμβιβαστικές τροπολογίες στο Συμβούλιο. Πιστεύω πως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για το συνολικό πακέτο όλων των τροπολογιών στις 23 Απριλίου, στον τέταρτο τριμερή διάλογο. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο Αναμένω τουλάχιστον θα μας κάνει μια λογική πρόταση. Κύριε Μάιερ, παρακαλώ, συνεδριάζουμε. Αν θέλετε να συζητήσετε ιδιωτικά με τα υπόλοιπα μέλη της γερμανικής αντιπροσωπείας, να το κάνετε έξω. Δουλέψαμε λοιπόν πάρα πολύ για τις εκτελεστικές και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. συμφωνήσαμε να συμπεριληφθούν στο ε, κύριο κείμενο ορισμένες από αυτές. Επίσης συμφωνήσαμε για πάρα πολλά τεχνικά σημεία. Υπάρχει βέβαια ένα κρεμές ζήτημα που αφορά την προέλευση των αγαθών στα τελωνία. Εκεί ακόμα πρέπει να συμφωνήσουμε για την ημερομηνία εφαρμογής. Και επίσης, εκ μέρους της κυρίας Λεγκρίπ, να σας ενημερώσω ότι επειδή δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μέχρι την ε, Ολομέλεια του Ιουλίου το νωρίτερο, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στον ε, ισχύον, στην ισχύουσα νομοθεσία για τα τελωνία και στην πρόταση. Προτάθηκε μία ξεχωριστή πρόταση που τροποποιεί την ισχύουσα εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά και να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα μέσα στο ισχύο νομικό πλαίσιο. Η κυρία Λεγκρύπ έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την συμπληρωματική νομοθεσία μαζί με τους κοιόδης εισηγητές. Τώρα, στις 2 Μαΐου θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σύσταση. Τα μέλη και οι συντονιστές θα λάβουν τις σχετικές πληροφορίες. Νομίζω είναι μόνο μία σελίδα νομοθετικού κειμένου. Και μετά θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας στον τριμερή διάλογο με στόχο να υιοθετηθεί όλο το πακέτο. Αυτά προς το παρόν για την έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ και τώρα νομίζω έχουμε ολοκληρώσει τις εκθέσεις. Αν υπάρχουν άλλα μέλη που έχουν σχόλια ή ερωτήσεις για αυτά τα σημεία, να το κάνουν τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εισηγητές και όσους εργάστηκαν για τους φακέλους αυτούς. Προχωράμε τώρα. Στο πρώτο σημείο θα συζητήσουμε την γνωμοδότηση της κυρίας Παρβανόβα για τα δικαιώματα των γυναικών ήταν κοινή πρόταση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την ισορροπία ανδρών και γυναικών για το ποσοστό των γυναικών στα μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη των εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η κυρία Χέντ δεν είναι εδώ, αλλά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ είμαι ο μόνος κοιόδης εισηγητής που βρίσκεται εδώ σήμερα το πρωί. Η κυρία Παρβανόβα και η κυρία Γκέμπχαρτ θα μιλήσουν για τους σοσιαλιστές. Έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία έγινε από κοινού με την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχουν πολλές ακόμα επιτροπές που ετοιμάζουν γνωμοδοτήσεις. Για την δική μας Επιτροπή είναι σημαντικό να δώσουμε λίγη σαφήνεια, διότι ο φάκελος είναι αρκετά περίπλοκος. Προωθείται λοιπόν η συμμετοχή των γυναικών στα μη εκτελεστικά διοικητικά ε, συμβούλια. Σύμφωνα με στοιχεία της ε, Κομισιόν, 15,8% των ε, θέσεων στις εταιρείες συγμένες στο χρηματιστήριο καταλαμβάνονται από γυναίκες και έχει παρατηρηθεί αύξηση 0,6% μόνο τον τελευταίο χρόνο εκτιμάται ότι οι γυναίκες ε, θα έχουν θετική συνεισφορά διότι οι γυναίκες αυτή την εποχή αποτελούν το 70% των καταναλωτικών δαπανών, των αποφάσεων για καταναλωτικές δαπάνες. Έχω ετοιμάσει τρει ομάδε τροπολογιών για τη δική μα επιτροπή. Η πρώτη έχει να κάνει με τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Περισσότερε γυναίκε σε διοικητικέ θέσει θα δώσουν μια ευρύτερη και σαφέστερη εικόνα τη ε, αγορά και θα τονώσουν τις πωλήσει. Επίσης, ε, από μελέτες έχει διαφανεί ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην ε, αύξηση των πωλήσεων και στη συμμετοχή των γυναικών. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών αφορά την ε, νομική σαφήνεια προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο σύστημα και η νομοθεσία είναι πολύ σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι οι εταιρείε που, που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά χρειάζονται ένα νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να ...εποφεληθούν από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά Και η τρίτη ομάδα τροπολογιών έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται γύρανση του πληθυσμού και γι' αυτό η μη επαρκή συμπερίληψη των γυναικών θα ε, έχει αρνητικές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, το γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό και εταιρείε πρέπει να έχουν κίνητρα για να συμπεριλαμβάνουν γυναίκες στα διοικητικά τους συμβούλια. Επίσης, η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 23 της Συνθήκης και να σας θυμίσω τέλος ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι την επόμενη Τετάρτη στις 17 του μήνα το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Good. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ο κύριος Ζουβέν θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Αλεγρή. Παρακαλώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, η κυρία Λεγρίπ που είναι η συγγήτρια για το Ελκ, μου ζήτησε να συνεισφέρω εκ μέρου τη. Καταρχήν ευχαριστώ την συγγήτρια για την γνωμοδότηση που προτείνει στην Κομισιόν. Το διάθεση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Καθώ το θέμα τη συμμετοχή ε, των γυναικών ε, στην λήψη αποφάσεων και κυρίω στα οικονομικά ζητήματα είναι πρωταρχική σημασία. Η κυρία Λεγκρίπ ε, συμφωνεί με τη γενική προσέγγιση που ακολουθεί η συγγήτρια, και υποστηρίζει το σχέδιο οδηγίας της Κομισιόν θα ήθελα να υπενθυμίσει ότι κατά την προηγούμενη τελική απόψη είχε την δυνατότητα να πει ότι έπρεπε να αλλάξει η νομοθεσία γιατί η αυτορύθμιση έδειξε τα ωριά τη. Πιστεύει ότι οι αριθμητικοί στόχοι θα είναι αποτελεσματικά εργαλεία βάσει τη εμπειρία που έχουμε σε πολλές χώρες. Ω εισηγητρία του ΕΛΚ μου ζήτησε να σα ενημερώσω ότι θα υποστηρίξει πολλέ από τις τροπολογίε της κυρίας Παρβάνοβα, κυρίως 2, 3, 5 και 9 Βέβαια, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Φαίνεται καταρχήν ότι κάποιε από τι τροπολογίε που έχουν να κάνουν με τα άρθρα τη οδηγία δεν είναι ε, παρκώ σαφεί από νομική αψή ή ίσω ε, δεν είναι καλή η μετάφραση και αναφέρεται συγκεκριμένα στα άρθρα 5 και 8 που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Κατόπιν, η κυρία Λεγκρίπ θέλει να υπενθυμίσει ότι εδώ και κάποια χρόνια άνω το 60% των ε, νέων πτυχιούχων ε, ε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς γυναίκες και ε, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του αριθμού των ανδρών και των γυναικών ε, στις διοικητικές ε, θέσεις που παραμένει αδικαιολόγητο και πρέπει να μειωθεί. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που θέλει να καταθέσει, αναφέρει τη δυνατότητα να εξεταστεί ο στόχος της οδηγίας να προσδιοριστεί το άρθρο 1 και πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως να σεβαστούμε τον ε, πολιτισμό, την κουλτούρα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και το δίκαιο των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά ε, το δίκαιο της επιχειρήσης. Επίσης, για το άρθρο 4-3 πιστεύει ότι θα πρέπει αυτά τα κριτήρια να είναι απολύτω ίσα για τι άνδρε και για τι γυναίκε. Επίση, αναρωτιέται σε σχέση με το τι θεωρεί η Κομισιόν ω το κατάλληλο στάδιο αυτή τη επιλογή για την εφαρμογή των διαδάξεων τη οδηγία και δεν απομακρύνει την δυνατότητα ε, να διασφαλιστεί η ευελιξία που θέλουμε σε σχέση με το δίκαιο των εταιριών. Επίσης, για την τροπολογία 6 ε, όπου αναφέρονται οι επιχειρήσεις ε, με λιγότερους ε, από 10 υπαλλήλου, Εκεί μου είπε να είμαστε υπέρ η κυρία Γκρίπ, όμως το θέμα αυτό συζητάται σε πολλές πολιτικές ομάδες. Για να κλείσουμε, η κυρία Γκρίπ ελπίζει ότι τις επόμενες εβδομάδες η συζήτηση με την κυρία Παρβάνοβα και τους σκιώδεις εισηγητές θα είναι επικοδομητική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τη συνάδελφό μου, διότι έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της. Είχαν ένα θάνατο στην οικογένεια και γι' αυτό μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω. Σήμερα όπως είπε και ο κύριος Ζουβάν και η κυρία Λεγκρίπ, έχουμε μια γενιά γυναικών που έχει άριστα προσόντα, όμως δεν έχει καμία πρόσβαση ή έστω πάρα πολύ χαμηλή πρόσβαση στις ε, πραγματικά αποφασιστικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι ενδεικτικό για το που βρίσκεται η κοινωνία μας σήμερα. Αν δεν αλλάξει κάτι δεν θα έχουμε καλή συνέχεια. Έπειτα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι όμιλοι, αλλά και όχι μόνο αυτοί, συνηθίζουν να συνδέουν την πρακτική αυτή με ένα πολύ στενέφασμένο πλέγμα που εμποδίζει τις γυναίκες να εισέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, έκθεση φυσικά της κυρίας Παρβανόβα, η οποία έχει δώσει μια πολύ καλή προσέγγιση και ακολουθεί μια πολύ σωστή ε, γραμμή. Στο σχέδιο έκθεσης τονίζονται οι διαφορές στους κανόνες περισσότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και τονίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, η συγγήτρια έχει την άποψη ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες, οι οποίοι να δίνουν ευελιξία στα κράτη-μέλη, να δώσουν τις λύσεις που πρέπει ανάλογα με την δική τους εθνική παράδοση και τα συστήματά τους. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τώρα, η κυρία Παρβανόβα στην τροπολογία 6 επιθυμεί μία εξαίρεση για τις επιχειρήσεις στις οποίες υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες με λιγότερο του 10%. Η εισηγήτρια πιστεύει πως αυτό πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά και να συζητηθούν και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτό. Η τροπολογία 9 τώρα δημιουργεί προβλήματα και αυτό είναι κάτι που με βρίσκει και εμένα σύμφωνη, διότι αναφέρεται η συνέπεια των επιχειρήσεων και η έλλειψη μάλλον της συνέπειας και η μη τήρηση ε, των κανόνων από τις επιχειρήσεις. Και εδώ χρειαζόταν συζήτηση. Τέλος, Υπάρχουν κάποια σημεία που η κυρία Χέτς και η ομάδα μας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά. Καταρχάς, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν ανοιχτοί και διάφανοι κανόνες για την πρόσληψη προσωπικού και στα εποπτικά συμβούλια των εταιριών. Διότι πολλές φορές οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται και κλεισμένων των θυρών και δεν υπάρχει κάποια δημοσιευμένη προκήρυξη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν πρέπει να γίνει πιο διάφανη και δωρεάν, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Επίσης, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, πρέπει πραγματικά να αναλογιστούμε εάν Η πρόταση αυτή θα αφορά μόνο τις, τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο και όχι όλες τις μεγάλες εταιρείες. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείε αυτές που είναι στο χρηματιστήριο να αποσυρθούν από αυτό για να μην τηρήσουν τους κανόνες, εάν αυτό γίνει υποχρεωτικό. Τέλος, όσον αφορά τις κυρώσεις, η κυρία Χέτς και η ομάδα μας πιστεύει ότι θα ήταν καλό οι κυρώσεις να είναι αυστηρότερες. Έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αναγκαστούν πραγματικά να τηρήσουν και να σεβαστούν τους κανόνες σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω πως έχει δίκιο. διότι αυτό μας δείχνει και η εμπειρία μας σε όλους τους τομείς όσον αφορά τις κυρώσεις και τις συνέπειες. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις της συναδέλφου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα, επειδή είμαι σκιώδη συζητητή για την ομάδα μου και δεν υπάρχει και κανένα άλλο εδώ από του πράσινου. Ξέρω ότι ε, ε η συνάδελφο Ρουλέ πρέπει να πάει πίσω στη Γερμανία λόγω οικογενειακών υποθέσεων. Η ανησυχία μου για αυτή την πρόταση είναι δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει πραγματικά το πρόβλημα. Χάρηκα ιδιαίτερως που η κυρία Παρβάνοβα έβαλε κάποιες τροπολογίες για το θέμα του να δίνει κανείς στις γυναίκες τη δυνατότητα να τις ενθαρρύνει να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις γιατί νομίζω ότι στο δημόσιο τομέα, η δική μου τουλάχιστον εμπειρία είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ε, ευθύνης ε, είτε πρόκειται για υπηρεσίες υγείας, είτε πρόκειται για δημόσια διοίκηση, είτε πρόκειται για εκπαίδευση αλλά σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες δεν βλέπουμε το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των γυναικών. Μου φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι πραγματικά το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την ότροπια και όπως λέει η κυρία Παρβάνοβα σε μία από τις τροπολογίες της, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μπορούν οι γυναίκες να αναπτύξουν όλες τους τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους ε, στην κοινωνία μας ε, κατά το μέγιστο δυνατό. Το πρόβλημά μου με αυτό και το έχω πει από την αρχή είναι ότι είναι μια ένα ιδιαίτερα επιλεκτικό μέτρο, το οποίο ουσιαστικά στοχεύει σε μία μόνο πτυχή και αφορά τα μη εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη. Το είπε και η κυρία Γκέπχαρτ. Δηλαδή, δεν θα στοχεύει στην ενθάρρυνση των γυναικών να λάβουν θέσεις ε, ε, εκτελεστικών διευθυντών, για παράδειγμα. Δεν λέω καλά, είναι και τα μη εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, γιατί μπορεί να ε, πιέσουν ε, τα υπόλοιπα μέλη ενός ε, συμβουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα καλύτερη υποβολή εκθέσεων, καλύτερες στατιστικές. Ξέρω ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις το κάνουν, το κάνουν ήδη σε μερικά κράτη-μέλη, σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη και αυτά τα ζητήματα. Το, το, η δική μου ανησυχία είναι και συμφωνώ Νομίζω ότι και η κυρία Γκέπχαρντ το υπονόησε στην τελευταία της παρατήρηση, είναι ότι το γεγονό ότι συνάδει κανεί με αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει, με αυτέ τι διατάξει, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η νοοτροπία τη επιχείρηση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πράγματι να συμβεί. Μπορεί να δώσουμε πολύ σημασία στη συμμόρφωση με τι νομικέ απαιτήσει ε, και την αποφυγή κυρώσεων. Όμω νομίζω ότι έτσι ουσιαστικά απομακρυνόμαστε από τι πραγματικέ ανησυχίε σε σχέση με αυτό το θέμα. Η δική μου ομάδα νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει βασική νομική λύση, αλλά θα κάνουμε σίγουρα συστάσεις για να μπορέσουμε τουλάχιστον να ασχοληθούμε με κάποια από τα ευρύτερα ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Όλοι συμφωνούμε με το πρόβλημα, αλλά δεν συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε για τη λύση του προβλήματο. Θα ήθελα να ενισχυθεί η διάταξη του άρθρου 8 που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που έχουν ήδη λάβει μέτρα να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη, πιο ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, να αναστείλουν ε, την εφαρμογή όλων αυτών των διαδικασιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για χώρες ε, σαν τη δικιά μου που ήδη ε, σημειώνουν ε, πρόοδο και νομίζω ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να πρέπει κανείς να εφαρμόσει μια πανευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, τη δημιουργία περίπλοκων συστημάτων προστήμων κλπ. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά απομακρύνει την προσοχή από την αντιμετώπιση του προβλήματος και πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην ενθάρρυνση τρόπων με τους οποίους οι εταιρείε αναπτύσσουν, εκπαιδεύουν, εμθαρρύνουν τις γυναίκες ε, να ανέβουν ε, ε, στην ιεραρχία της εταιρείας τους. Της εταιρείας τους. Θα ήθελα πιο πολλούς εκτελεστικούς διευθυντές. Γιατί αυτοί είναι που θα αλλάξουν την πραγματική νοοτροπία των εταιριών. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες συστάσεις στην κυρία Παρβάνοβα και ελπίζω να σημειώσουμε πρόοδο. Στάιλερ και Κρόιτσμαν. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. κυρία Βερχάιν. Κυρία ε, Στάιλερ πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Παρβανόβα για την έκθεση. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία για το πόσο συχνά ε, πόσο χαμηλά μάλλον ε, χαμηλώνει το ποσοστό των γυναικών και πόσο χαμηλή η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στις ηγετικές θέσεις. 6% ε, νομίζω αναφέρεται. Είναι πολύ χαμηλό. Εμείς θέλουμε αύξηση κάθε χρόνο και πρέπει να αναλάβουμε δράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σχολή ε, δημόσιας διοίκησης ε, ε, αναφέρθηκε σε μια έκθεση που έχει να κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο και στο πρώτο ημίση του οικονομικού έτους υπήρχε μια αύξηση 44% και το δεύτερο εξάμεινο μόνο 26%. Και η έκθεση λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει συνενοχή των εταιριών. Ε, επειδή δηλαδή στο πρώτο εξάμεινο υπήρχε κάλυψη του θέματο από τα ΜΜΕ ε, ανέλαβαν μεγαλύτερη δράση, ενώ το δεύτερο εξάμεινο φυσικάστηκαν. Και έτσι λοιπόν ανθίστανται οι εταιρείε ε, στο να κάνουν σημαντικέ αλλαγέ, Αναφέρθηκε στην αλλαγή της κουλτούρας ε, ο πρόεδρος. Μερικές φορέ είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο από διάφορου οργανισμούς και βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι γυναίκες καλύπτουν μόνο το 17% των θέσεων, πολύ πιο κάτω από το στόχο τη κυβέρνηση, που είναι το 25% και από τις 250 εταιρείε, μόνο το 27% αυτών των εταιρείων έχουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και ξέρουμε ότι οι γυναίκες έχουν ταλέντο και ικανότητες και μιλάμε για το 70% ε, του πληθυσμού. Οι γυναίκες αποτελούν το 70% ε, του πληθυσμού και έτσι λοιπόν ε, υπάρχει λόγος να έχουμε και εκπροσώπηση γυναικών στις εταιρείες. Αν δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ναι, ε, για την ε, ποιότητα. Επίσης ε, πρέπει να δούμε και τι είπε η έκθεση. Δεν νομίζω ότι τα εθελούσια μέτρια λειτουργούν. Εγώ είμαι υπέρ των ποσοστώσεων στα συμβούλια. Ξέρω ότι κάποιοι δεν το θέλουν, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε ισορροπία εκπροσώπησης των δύο φύλων στα συμβούλια πριν να φτάσω τα 100. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν και πάρα πολύ πολύπλοκα θέματα για την οικογενειακή ζωή, για τη φροντίδα των παιδιών, για το περιβαλλον εργασίας, για το πώς θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους ε, να ακολουθήσουν κάποια σταδιοδρομία και να υπάρχει υποστήριξη και όλα αυτά. Όμως, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται δράση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Συμφωνώ, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση. Είπα ότι αυτό το μέσο δεν μας ε, διευκολύνει. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Καταρχάς πρέπει να διαχωρίσουμε τα εποπτικά από τα μη από τα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντούχες οι γυναίκες με εξαιρετικά προσόντα, οι οποίες θα ήταν πιο εύκολο να μπουν σε κάποια εποπτικά συμβούλια. Δεν ξέρω, το κόμμα μου είναι κάπως σκεπτικό όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Επίσης η κυρία Γκέμπχερτ πρέπει να λάβει υπόψη της στις συζητήσεις στη Γερμανία διότι δεν υπάρχουν μόνο τα εποπτικά συμβούλια, υπάρχουν και τα συνδικάτα και εκεί πρέπει να εφαρμοστούν λοιπόν ποσοστώσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι σοσιαλδημοκράτες συνάδελφοι. Τώρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε επίπεδο προέδρων. Ναι, εκεί φυσικά και χρειάζονται οι γυναίκες με προσόντα, αλλά χρειάζεται χρόνος. Δεν θα γίνει από σήμερα μέχρι αύριο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις πρακτικές τόσο γρήγορα. Και αυτό θα ήθελα να πω. Ότι οι γυναίκες έχουν επίσης το πρόβλημα είναι ας πούμε σε μια μειονεκτική θέση επειδή κάποια στιγμή κάνουν παιδιά και μένουν εκτός. Και όταν είσαι σε μια ηγετική θέση ως γυναίκα πρέπει να κάνεις ορισμένες επιλογές υπέρ της καριέρας και όχι υπέρ της οικογένειας. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές, υπάρχουν διαφορές σε κλάδους, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους χρειάζονται περισσότερες γυναίκες και υπάρχουν επίσης κλάδοι όπως τεχνική κλάδη για παράδειγμα όπου υπάρχουν διαφορές και σε εκείνους τους τομείς χρειάζεται χρόνος έτσι ώστε να μην γίνουν λάθος βήματα και λάθος ε, σπασμωδικές κινήσεις. Πρέπει να ε, διεξαχθεί λοιπόν ομαλά αυτή η μετάβαση. Γι' αυτό πιστεύω πως αυτό δεν έχει να κάνει με τα δίκτυα που αναφέρατε. Για παράδειγμα, το θέμα των παιδιών, των γυναικών και των παιδιών, το έχουν καταλάβει πλέον οι μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχουν λύσεις γι' αυτό, υπάρχουν οι παιδικοί σταθμοί. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις ποτέ δεν θα προσλάβουν σε υψηλή θέση μια γυναίκα η οποία έχει παιδιά και η οποία πρέπει να τα αφήνει κάθε μέρα στον παιδικό σταθμό και να αναγκάζεται να τα αποχωρίζετε όλη την ημέρα. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι λοιπόν τόσο πολύ ποσοστώσεις, αλλά πρέπει να αποδομήσουμε αυτή τη μειονεκτική θέση. Όπως είπατε, να αλλάξει η νοοτροπία. Αλλά αυτό όμως πρέπει να γίνει σιγά και πρέπει να γίνει με τις σωστές προϋποθέσεις. Εάν δεν υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις, τότε οι γυναίκες πάντα θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Δεν θα αλλάξει αυτό. Uh, thank Σας ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν. Να ακούσουμε την κυρία Βαχένα και με την ε, κυρία Πέρες. Κυρία Βαχέν, καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί είναι αντιφατικά. Όπως είπα και ο κύριος Κρότσμαν, στη τελική ανάλυση πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να μην βιαστούμε. Το να βάλουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει οι επιχειρήσεις να υφετήσουν αυτές τις ποσοστώσεις, δεν θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να υπάρχει χρόνος, πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε η αλλαγή να γίνει σε βάθος χρόνου και να γίνει μόνιμη. Πόσο θα χρειαστούμε, 10, 15, 20 χρόνια. Συζητάτε αυτό το θέμα για την, ε, την μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, υψηλέ θέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν προσόντα, οι οποίες κατάφεραν να ανέβουν ψηλά στην σκάλα των συμβουλίων αυτών, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται και σε ιδιαίτερα τεχνικής φύσης θέση. Και όπως είπατε, υπάρχει και το, μεγάλο το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, αποφύτων στις ε, τεχνικές σχολές είναι γυναίκες πλέον. Πραγματικά, όμως, Κύριε Κρόιτσμαν, εσύ που αναφέρατε το θέμα των ε, παιδιών, δεν ξέρω αν αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δεν νομίζω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δημιουργική συζήτηση. Και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, πραγματικά. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, οι ποσοστώσεις δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως ένα πρώτο βήμα. Έτσι ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες στις θέσεις των διοικητικών συμβουλίων. Χρειάζονται υποδομές. Όπως είπαμε, χρειάζονται πιο ευέλικτα ωράρια, χρειάζονται χρειάζονται παιδική σταθμή, χρειάζονται προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν τις γυναίκες μακροπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η κυρία Πέρες. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες ε, παρατηρήσεις κατόπιν των όσων ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες ε, και θα ήθελα να αναφερθώ και στα επιχειρήματα της κυρίας Τάιλερ. Κατανοώ ότι όλοι οι συνάδελφοι που βρισκόμαστε εδώ είμαστε άνθρωποι του καιρού μας. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ έναν Ισπανό φιλόσοφο, τον Ορτέγα Γασέρ, ο οποίος είπε ότι ο άντρας ή η γυναίκα που δεν συνάδει με την εποχή του ουσιαστικά δεν ζει τη ζωή του όπως πρέπει. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιούμε το τι βιώνουμε και σήμερα ε, οι γυναίκες αποτελούμε πάνω από το 50% του πληθυσμού και είμαστε σε υποκροσώπηση σε ό,τι αφορά τις ε, υψηλές διοικητικές θέσεις. Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα για τις γυναίκες, όμως δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί εμείς είμαστε ικανές ως γυναίκες να κάνουμε διάφορα πράγματα και πέρα από το ότι είμαστε ικανές, έχουμε και τα κατάλληλα προσόντα και θα πρέπει να πάμε στο σύστημα των ποσοστώσεων, γιατί ξέρουμε ότι κοστίζει ε, πάρα πολύ. Τώρα προχωρήσουμε έτσι λοιπόν όταν ε, δεν σημειώνεται πρόοδο, τελικά σημειώνεται η παναχώρηση. Όπω ε, είπε και ο Πρόεδρος, πέρα από το άρθρο 8 πρέπει να πάμε. Ναι, να έχουμε παιδικού σταθμού, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και τη σημερινή κουλτούρα που επικρατεί, που δεν αντιμετωπίζει τι γυναίκε ω ισότιμε. Σα ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Είχαμε ευρία συζήτηση μέχρι τώρα. Θέλει κάποιο άλλο να συνεισφέρει. Νομίζω ότι έχουμε και εκπρόσωπο της Κομισιόν. Επομένως, ε, δεν έχει προγραμματιστεί βέβαια. Θέλετε όμως το λόγο, Μιχαήλ Γκάντε. Είμαι νομικός εκπρόσωπος στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνης, στην, αρμόδια μονάδα για την ισότητα των δύο φύλων. Δεν έχουμε συγκεκριμένα σχόλια για τις τροπολογίες, όμως εκ μέρους της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια για το έργο της και την Επιτροπή για ότι εργάστηκε ταχύτατα για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή θέλει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στα κράτη-μέλη για τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν σας ευχαριστούμε γιατί έχετε εργαστεί ταχύτατα για το του αυτού μέχρι σήμερα. Κυρία Παρβάνοβα, θέλετε να, συνο... συνοψίσετε και να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις και όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα είναι δύσκολο να, την, να αλλάξουμε την κουλτούρα στις εταιρείε, όμως ε, από ό,τι φαίνεται από τα δεδομένα τα τελευταί, τους τελευταίους δύο αιώνες δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο με φυσικό τρόπο. Έτσι λοιπόν ίσως ήρθε η στιγμή να νομοθετήσουμε και Είμαστε πάρα πολύ περηφανοί επειδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η ηγετική δύναμη παγκοσμίω για την ε, επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων γυναικών. Επομένω, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα να νομοθετήσουμε ε, όχι μόνο για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, αλλά ίσω και στην πολιτική. Λοιπόν, για να μπούμε σε φιλοσοφική συζήτηση, θα έλεγα ότι θα βάλω τα δυνατά μου για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για τα συμφέροντα της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και λαμβάνοντας υπόψη της θέσης της ΣΥΜΚΟ και είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την τροπολογία 6 για ε, αν, αν υπάρχει ε, κάτω από το 10% του εργατικού δυναμικού ε, των εταιριών, αν οι υπάλληλοι δηλαδή που υπεκρισωπούνται, το φίλο που υπεκρισωπούνται είναι κάτω από το 10% του εργατικού δυναμικού, δεν έχει σημασία γιατί ε, επίσης ε, έχει αποδεικτεί ότι ε, για τις επιχειρησιακές ε, λειτουργίες ε, δεν θα έπρεπε να θέτει πρόβλημα το θέμα του φύλου. Και έχουμε εταιρείες στις οποίες υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. επειδή υπάρχουν μικρότερες ευκαιρίες να μπουν σε αυτούς τους τομείς το χάρη όταν μιλάμε για τον τραπεζικό τομέα και το τομέα των ασύμων πηγών ενέργεια. Για μια ακόμη φορά θα αναφέρω το χρονοδιάγραμμα και ανυπομονώ να λάβω τις τροπολογίες. Και θα έχουμε μία συνάντηση των σκιωδών και θα συμφωνήσουμε για το ποια θέση θα είναι κατάλληλη να υιοθετήσουμε ως 17 Απριλίου το μεσημέρι προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. έχει προβλεφθεί για τις 29 Μαΐου και κατόπιν 30 Μαΐου η ημερομηνία έγκρισης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Παρβάνοβα για τη δουλειά αυτή και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Καλύψαμε αυτό το θέμα στο χρονικό περιθώριο που είχαμε και να περάσουμε τώρα στις δύο ψηφοφορίες για σήμερα. Πρώτον, έχουμε τη γνωμοδότηση για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ευεργέτημα παινία σε διασυνοριακές πολιτικές και εμπορικέ ε, διαφορές. Hans Peter Mayer. Να του δώσω λίγο το λόγο να μας κάνει μια εισαγωγή και να πει ορισμένα πράγματα και αν δεν θέλει μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Θέλετε να μας πείτε ορισμένα πράγματα, κύριε Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι να σας μοιραστεί λοιπόν ο κατάλογος της ψηφοφορίας, να πω ότι το θέμα είναι αρκετά δύσκολο. Υπάρχουν διασυνοριακές διαφορές και το πρόβλημα είναι τι γίνεται σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν έχουν χρήματα για εκπροσώπηση. Έχουμε καταλήξει σε ορισμένους συμβιβασμούς στον κατάλογο. Υπάρχουν μία-δύο προφορικές τροπολογίες. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα ε, με αυτές, όπως ε, μας ενημέρωσαν και οι υπόλοιπε ομάδες. Έτσι πιστεύω πως όλα θα εξελιχθούν ομαλά για το καλό των πολιτών. Ευχαριστώ. Right. Ωραία. Θέλει κανείς από τους σκιώδει ηγητέ να πάρει το λόγο? Ωραία, α περάσουμε τότε στην ψηφοφορία. Θα αρχίσω με την τροπολογία 1. Νέα παράγραφος από τον εισηγητή υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 κυρία Πέρες υπέρ κατά. Αν έχετε όλοι τις κάρτες σας, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 3. Εγκρίνεται. 13-7. Πρώτη συμβιβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την 7 της κυρίας Πέρες. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα εδώ, οπότε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ο κύριος Ζιβάν δεν έχει την κάρτα του. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 12 κατά. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 8, 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 με, προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Δύο τμήματα. Το ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, 17 λοιπόν. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18. Ιριγκόιεν Πέρες. Υπέρ. Ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 18. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-16. Τροπολογία 19. Μάιερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20. Ριγόιεν Πέρες. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός και για αυτήν. Πέρας. Της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 11-17. 21. Πέρες, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση του κυρίου Μάιερ. Ανεβαίνουν οι αριθμοί. Πέρας. Εγκρίνεται 27 υπέρ. Κανείς κατά και μία αποχή. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάιερ. Θα επερασπιστείτε έτσι τη θέση μας στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας για τα είδη πυροτεχνίας. Ένα, μία, μία ψηφοφορία θα κάνουμε για την αποδοχή του αποτελέσματος της ε, συνδιαλλαγής. Να δώσω όμως το λόγο στην εισηγήτρια να μας πει ορισμένα πράγματα, να μας ενημερώσει κάπως για το πώς έχουν τα πράγματα για το υπόλοιπο νομοθετικό πακέτο και τις συναντήσεις του τριμερούς διαλόγου. Να σας δώσω λοιπόν το λόγο, κυρία Ροϊτόβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω απλώς ότι ο τριμερής διάλογος αφορούσε το ένα τμήμα ε, του πακέτου εννέα ζητημάτων. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έχουν αρχίσει από τον Νοέμβριο και πρέπει να πω ότι αυτή η οδηγία Ε, την ξεχωρίσαμε κάπως και την προωθήσαμε γιατί ήταν σημαντικό η ε, ενημέρωση να γίνει πριν από τον Ιούλιο ε, και την δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα με τους αερόσακους των αυτοκινήτων. Ήταν δυνατό να υπερασπιστούμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες μας θα εξυγχρονιστούν οι κανόνες και επομένως ε, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να οργανώσουν ε, την ε, παραγωγική τους διαδικασία καλύτερα και θα μπορέσουν να τοποθετήσουν τα σχετικά προϊόντα στην αγορά πολύ πιο γρήγορα. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλέστερα προϊόντα και αυτό γιατί οι εποπτικές αρχές θα έχουν περισσότερες εξουσίες να αποσύρουν επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά και να επιβάλλουν κυρώσεις ε, στους εισαγωγείς, ειδικότερα αν ε, υπάρχουν προϊόντα κακής ποιότητας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, γιατί θα υπάρχει ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας ε, των ειδών πυροτεχνίας, θα υπάρχουν θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ε, απαραίτητα στοιχεία, κάτι το οποίο θα είναι ευκολότερο στην πρόσβαση για τον καταναλωτή. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις και με την Κυπριακή και με την Ιρλανδική Προεδρία ήταν πάρα πολύ καλές, όμως προς το τέλος προέκυψε το θέμα του ρόλου των κρατών μελών στην επιτροπολογία. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από την έλλειψη εμπιστοσύνης των κρατών μελών εδώ και κάποια χρόνια, πέρα από το πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας, προσπαθούσαν, προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε τους ε, εμπειρογνώμονες των κρατών μελών να συμμετέχουν απευθείας στις διαπραγματεύσεις, όμως ε, αυτό δεν είναι ε, κατά την αυστηρή έννοια του όρου δεν προβλέπεται στο συγκεκριμένο πακέτο. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις, όμως κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο, με πολλή βοήθεια από τον πρόεδρό μας, προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή διατύπωση ε, ώστε να είμαστε σε συμφωνία και με το Συμβούλιο κυρίως για το πρωτογενέ δίκαιο μιλάω, υπήρξε με ένα συμβιβασμό ε, για, στην Κορεπέρ, εκτός από το κομμάτι αυτό που αφορά την, αφορά την επιτροπολογία. Αντί για standard, standard rules of procedure, μιλάμε για rules of procedure of the relevant committee. Τους κανόνες δηλαδή της αρμόδιας επιτροπής όλα τα δέχτηκε η Κορεπέρ, εκτός από αυτό το σημείο το οποίο άλλαξε όπως σας εξήγησα. Δεν είναι τεράστια διαφορά και κανονικά οι γλωσσομαθείς νομικοί θα ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Ελπίζουμε όμως ε, ότι και το Συμβούλιο και εμείς θα εγκρίνουμε το σχετικό έγγραφο. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη Μαΐου να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να μην προβαίνει σε τέτοιου είδους αλλαγές τελευταία στιγμής, γιατί δεν απαιτείται κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του πακέτου. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να γίνει τέτοιου είδους ε, ε τελευταία στιγμής προσαρμογή και δεν θέλουμε να υπάρξουν εμπόδια στην ολοκλήρωση 8 οδηγιών πριν από τις καλοκαιρινές ε, διακοπές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας. Να ευχαριστήσω ε, τους ε, τους κοιόδης εισηγητές, τους βοηθούς μου, το προσωπικό της Επιτροπής μας. Ήταν όλοι πάρα πολύ ευέλικτοι. Καταφέραμε να βρούμε τις σωστές αποχρώσεις στο κείμενο για να διατηρήσουμε τη θέση που είχε εγκρίνει η Επιτροπή μας και επίσης ε, καταφέραμε να καταστήσουμε το κείμενο αποδεκτό και για τους εταίρους μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω ε, να υπερψηφίσετε ε, την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς από τους σκιώδεις εισηγητές να πάρει το λόγο? όχι. Ωραία. Τότε θα κάνουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα πρακτικά Αρχίζουμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία για ε, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής για την αγορά ειδών πυροτεχνίας. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται 28 υπέρ. Καμία ψήφος ε, κατά και μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρόιτοβα. Οπότε αυτό το πακέτο θα είναι τμήμα της ημερήσιας διάταξης ε, της Ολομέλειας του Μαΐου θα υποβληθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι όπως είπε και η κυρία Ρόιτοβα είναι μια πολύ καλή βάση για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο πακέτο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε θα συνεχίσουμε του τριμερού διαλόγους ε, το Μάιο για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό με το Συμβούλιο γιατί καταφέραμε να λύσουμε ορισμένα ζητήματα για τις εκτελεστικές και τις κατεξιοδότης πράξεις. Υπήρξε πολύ τεχνική δουλειά που έγινε και η Σουζάν συμμετείχε και εκείνη, ε, η δική σου ομάδα, η βοηθή σου, Νομίζω ότι ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόση πολλή δουλειά γίνεται για τις λεπτομέρειες ενός τέτοιου είδους ε, θεμάτων, ενός τέτοιου θέματος, οπότε θα ήθελα να το πω αυτό και για τα πρακτικά. Ελπίζω να έχουμε ένα ευθυγραμμισμένο κείμενο με το Συμβούλιο, ώστε να μην αποδεχθούμε απλώς αυτό που θέλει το Συμβούλιο χωρίς να το εξετάσουμε κι εμείς. Περνάμε τώρα σε πρόταση ψηφίσματος για τις τροπολογίες της πρότασης Τη Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το εμπόριο και τις επενδύσει. Αν θυμάστε, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μας κάλεσε να υποβάλουμε ορισμένε τροπολογίε ή προσθήκες. Αυτό το διαχειρίστηκαν οι πολιτικές ομάδες και είχαμε πολλέ ευκαιρίε να το συζητήσουμε. Τώρα λοιπόν υποβάλλεται προσέγγιση. Δεν έχουμε εισηγητή ε, δεν ξέρω αν κάποιο από του εισηγητέ των πολιτικών ομάδων θέλει να σχολιάσει, αν προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ίσως στο μέλλον θα έπρεπε να ορίσουμε κάποιον μόνιμο εισηγητή για τι εμπορικέ διαπραγματεύσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό θα το συζητήσουμε στου συντονιστέ. Πιστεύω πω θα ήταν καλή ιδέα για το μέλλον. Και να έχουμε κάποιον συντονιστή ο οποίος θα εναλλάσσεται ένα πολιτική ομάδα. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τις τροπολογίες. Λοιπόν, αρχίζουμε με την παράγραφο 2, τροπολογία 13 του κυρίου Βάιντεν Χόλτσερ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 14 αποσύρεται. 15 του κυρίου Λόκεγκαρτ υπέρ. Ποιο είναι κατά. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 21 της κυρίας Γκάλιο. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 20 κυρίου Βάιντενχόλτσερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 22. Σάλτε Μούζε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 του κυρίου Τρασκόφσκι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας εμένα. Εγκρίνεται η τροπολογία μου. 27 της κυρίας Φερχάιεν υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. 28 της κυρίας Κοράτσα Μπίλ και λοιπόν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 29 του κυρίου Βάιντεν Χόλτσερ, ποιος είναι υπέρ, ποιος κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 30, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, δική μου, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 32. Με προφορική τροπολογία του κυρίου Σφάμπ και άλλων. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 του κυρίου Σφάμπ και άλλων. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 35 ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 39 είναι χωριστή ψηφοφορία, όπως ζήτησαν οι ελεύθεροι. Πρώτο μέρος λοιπόν, ποιος είναι υπέρ, ποιος κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 40, ποιος είναι υπέρ, ποιος κατά, εγκρίνεται. 41, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 συνδέεται με τη 18, άρα εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Λόκεγκαρτ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 έχει μια προσθήκη τη λέξη consumer, καταναλωτή υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. να δούμε τις 9, 10, 11 και 12 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Απορρίπτονται όλες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα τις καταθέσουμε ως σύνολο στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και προς πληροφόρησή σας η ψηφοφορία στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι στις 24 και 25 Απριλίου. Θα ψηφίσουν στην Ολομέλεια του Μαΐου. Κύριε Σφάμπ, θα θέλατε κάτι? Όχι. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει ίσως κάποιος από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ολοκληρώνει την ψηφοφορία μας για σήμερα. Περνάμε τώρα Έχουμε κερδίσει και τρία λεπτά. Αν συμφωνεί ο συγητής λοιπόν θα προχωρήσουμε αμέσως. Όποιο θέλει να φύγει τώρα μπορεί να φύγει παρακαλώ ήσυχα όμως για να συνεχίσουμε εμείς τις εργασίες μας. Τώρα λοιπόν θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ντεκάμπος για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή τον καθηγητή Ντεκάμπος. Έπειτα θα πάρει το λόγο ο κύριος Σβάμπ, ο κύριος Μπίλαν και ο κύριος Μέντες. Ίσως και κάποιος από τους πρασίνους. Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε κάποιον από τους πρασίνους. Το λόγο έχουν σκιώδεις εισηγητές λοιπόν και όποιος άλλος θα ήθελε. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή. Δεν νομίζω. Αν έρθει κάποιος, νομίζω θα είναι η κυρία Μπερνάρ. Δεν ξέρω αν πληροφορήθηκαν για την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε εκπονήσει μια γνωμοδότηση υπόψη του κυρίου Μποζέκα για το πώς θα λειτουργήσει η εσωτερική αγορά ενέργειας. Έχουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας που βρίσκεται στην αρχή της. Έχουμε πάρα πολλά εμπόδια που παραμένουν και λείπει μια ολοκλήρωση που να μεταφραστεί σε ανταγωνιστικότητα έτσι ώστε να φτάσουμε στη μείωση των τιμών και στην επίτευξη άλλων ε, και άλλων πλεονεκτημάτων για τον, για τον καταναλωτή. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο δεν έχει μεταφερθεί ακόμη ούτε καν σωστά στην ιστορική νομοθεσία των κρατών μελών και υπάρχουν ε, κάποιες ε, κυρώσεις που προβλέπονται για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μεταφέρει την νομοθεσία στο ιστορικό της δίκαιο. Πρέπει να διακοπούν ε, οι επιδοτήσεις που διαστρεβλώνουν την αγορά, όπως επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και να εισαγάγουμε συνοχή για την υποστήριξη, για τη στήριξη των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, πρέπει να εφαρμοστούν διδάξεις του μηχανισμού για τη σύνδεση της Ευρώπης. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα προγράμματα που έχουν αμεσότερες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα την ένταξη των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειων, των ανταγωνισμών, ε, τη διαχείριση της ενέργειας ενέργεια και την ασφάλεια φοδιασμού. Πρέπει επίση να ε, βελτιώσουμε τα ωφέλη για τον καταναλωτή και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ενέργειας να υπάρχει προστασία των καταναλωτών, των πλέον ευάλωτων και συνεχής ενημέρωση νέος μηχανισμός για την επίλυση των διαφορών ε, μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών είναι κάτι απαραίτητο. Επίσης πρέπει να προωθηθούν μηχανισμοί και πρωτοβουλίε για να συμμετέχουν πιο ενεργά οι καταναλωτές στην ιστορική αγορά ενέργειας και ταυτόχρονα να υποφελούνται. Πέρα από τις πτυχές αυτές υπάρχουν και άλλες πτυχές που θέλουν να συμπεριληφθούν στην ε, νομοδότηση όπως να εφαρμοστούν γρήγορα κωδικοί δικτύου, για ε, να υπάρχει ολοκλήρωση των εθνικών αγορών. Όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε έτσι καλύτερη ροή της ενέργειας ε, στην αγορά και θα έχουμε καλύτερο ανταγωνισμό και περισσότερο ανταγωνισμό. Θα ήθελα να κλείσω χαιρετίζοντας όλους και όλες τις συναδέλφους ε, που βοήθησαν, που συνέβαλαν και με τη συμμετοχή όλων μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που παρουσιάζει τις διάφορες ανησυχίες αυτής της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο ρόλος μας εδώ είναι πέρα από το να βρούμε τις κύριε, τέλειες τεχνικές λύσεις να υπερασπίσουμε τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θέλει μια ξεκάθαρη λειτουργία της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκάμπος για την γνωμοδότηση, διότι πιστεύω ότι ήταν σύντομη και σαφέστατη. Χρειάζεται μία αλλαγή, λοιπόν, στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Εμένα... Και εμένα μου αρέσει και η πρώτη πρόταση και η δεύτερη για την εφαρμογή διότι πιστεύω πως η εφαρμογή και η αλληλεγγύη είναι η κύρια προτεραιότητα και πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να πιέσει η Κομισιόν τα κράτη-μέλη για να κάνουν τις αλλαγές αυτές. Φυσικά και χρειαζόμαστε αυτές τις ε, διασυνοριακές υποδομές, διότι αν δεν υπάρχουν αυτοί δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και η εσωτερική αγορά. Και αυτά που θα αποφασίσουμε εμείς εδώ δεν θα έχουν καμία απολύτως πρακτική εφαρμογή. Τώρα όσον αφορά το ρύθμιση των τιμών στην οποία αναφέρατε, αυτό είναι μεν αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως πιστεύω πως θα μπορούν να γίνουν, να γίνουν μερικές προσθήκες. Για παράδειγμα, μια καλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις ε, παραβιάσεις των, ε, στις διαδικασίες επιπαραβάσης των ε, κρατών μελών διότι είναι σαφές πως τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει υποχρεώσεις και από την άλλη υπάρχει και η εφαρμογή του ε, δικαίου περί κανόνων ανταγωνισμού, το οποίο, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να το τηρήσουν. Έπειτα, θα μπορούσε να γίνει σαφέστερη η αναφορά στα δικαιώματα και στις ε, στους εκλάδους ε, οι οποίοι θα πρέπει να υποστούν μέχρι το 2017. Επίσης, για να καταφέρουμε από το 2014 και μετά να επιτύχουμε μια καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να γίνουν καινούργιες διαδικασίες. Τώρα όσον αφορά την Βουλγαρία και την Ρουμανία και εκεί χρειάζεται να γίνουν νέες ενέργειες όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και τους παρόχους ενέργειας πρέπει να γίνουν συμφωνίες ή να συσταθούν εκ νέου συμφωνίες για την εσωτερική αγορά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε Τεκάμπος, θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω δύο σημεία τα οποία εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά αυτή η έκθεση για μένα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω πως πραγματικά κινδυνεύουμε στην Ευρώπη να στερέψουμε από ενέργεια, να έχουμε πρόβλημα. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Τώρα για τα επίπεδα προστασία αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε διότι το θέμα τη προστασία των καταναλωτών δεν αφορά μόνο την ε, παροχή ενέργεια. υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί κανόνες που διέπουν διάφορους τομείς και πιστεύω πως αυτοί πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Έπειτα, το αίτημα για την δημιουργία νέων μηχανισμών επίλυσης ε, διαφορών είναι πραγματικά Πάρα πολύ καλό και το χαιρετίζω. Επίσης, ε, χαιρετίζω και την πρόταση για εναλλακτικέ μεθόδους επίλυσης διαφορών. Πρέπει όμως να προσέξουμε αυτοί οι δύο μηχανισμοί να συσταθούν έτσι ε, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και σε συνεργασία. Τέλος, να ευχαριστήσω όλους σας και πιστεύω πως έχουμε καταλήξει σε ένα μια καλή πρόταση και συμβιβασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μάντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για τις προτάσεις της. Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν αλλαγές στην εσωτερική αγορά όσον αφορά την ενέργεια. Τώρα για τη σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα συνθήματα. Πιστεύω καταρχάς ότι πρέπει να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Έπειτα, αν δούμε την ενεργειακή εσωτερική αγορά, θα δούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν οι σωστές υποδομές για ηλεκτρισμό, για ηλεκτροδότηση και να υπάρχουν επενδυτές, θεσμικοί επενδυτές, διότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω ακούσει ότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ Ολλανδικά αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένα στο Λουξεμβούργο. Εάν λοιπόν οι φορείς αυτοί αποσύρουν αυτά τα 3 δισεκατομμύρια και τα επενδύσουν, τότε θα έχουμε καλύτερη απόδοση. Θα ωφελήσει όλους για παράδειγμα, θα ωφελήσει πάρα πολύ ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις ανεμογεννήτριες. Αν δημιουργηθεί ένα σωστό δίκτυο, τότε θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε και την ενέργεια. Έχουμε τα μέσα και ο κύριος Μπαρόζο μίλησε για το 2020 και είπε ότι μέχρι το 2020 ο μηχανισμός αυτός θα έχει τεθεί σε ισχύ. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει επιτέλους το πρόβλημα της ε, ενεργειακής έλλειψης και όσον αφορά ε, την στρέβλωση της αγοράς. Είναι πολύ εύκολο να προχωρήσουμε σε απελευθέρωση της αγοράς, είναι πολύ δύσκολο όμως αυτό να γίνει με τρόπο ώστε η αγορά να λειτουργεί με δίκαιο και σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω σε μια σωστή και θετική συνεργασία και πιστεύω πως θα βοηθήσει όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Νταμπίλιαν, είναι η τελική σκιώδη συγχύτρια και μετά η κυρία Στάιλερ θα λάβει το λόγο και όποιος άλλος θέλει. Κύριε Πίλερ. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκάμπος για την γνωμοδότησή του και να καλωσορίσω ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης γιατί είναι ο τελικός καταναλωτής ο οποίος πληρώνει τελικά για την ε, αναλοκληρωτή αγορά ενέργειας. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο αν είναι αρκετά ανταγωνιστική αγορά από τη σκοπιά του καταναλωτή σε ορισμένα κράτη-μέλη εξακολουθεί να είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς πάροχο ενέργειας. Ε, κάποιοι καταναλωτές ούτε καν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και το θέμα του ανοιχτού ανταγωνισμού και της ε, μη εισαγωγή διακρίσεων ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις υποδομές είναι επίσης κάτι ζωτικό για να αναπτυχθεί περαιτέρω η ενεργειακή αγορά η αποτελεσματική κρίση των υφιστάμενων δικτύων έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους ε, στην τιμή της ενέργειας είναι σημαντικό και τα φύ δίκτυα είναι κάτι σημαντικό επίσης. Όλα αυτά πρέπει να τονιστούν στη γνωμοδότηση. Πέραν όλων όσων υπάρχουν ε, ό,τι αφορά τα νομοθετήματα, σε επίπεδο νομοθετημάτων. η ολιστική προσέγγιση στην ε, ανάπτυξη της ε, αγοράς ε, ενέργειας είναι κάτι που θα συνεισφέρει στο να αναπτυχθεί καλύτερα η αγορά. Εγώ θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και για αυτή την ευκαιρία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τους Κιώδης. Ας ε, ανοίξουμε τη συζήτηση με την κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντική η έμφαση που δίνεται στην παράγραφο 5 σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές ε, καθώς ε, το κόστος των καυσίμων για πολλές οικογένειες αυξάνεται και δημιουργεί πολύ μεγάλες πιέσεις για τα νοικοκυριά και Επίσης, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, πρόσφατα είχαμε κατάχρηση της πωλήσει ε, και το θέμα είναι πώς οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν πάροχο και να ενημερωθούν γι' αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία για το community switching. Ε, δεν ξέρω αν ο εισηγητή ε, γνωρίζει αυτό το θέμα και αν υπάρχουν ε, βελτιστέ πρακτικές που μπορούμε να ανταλλάξουμε για τέτοιε πρωτοβουλίε Είναι πολύ σημαντικές. Ε, και όπως ε, είπα υπάρχει πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά και η ενεργειακή ανέχεια είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι είχαμε και έναν από τους ε, πιο κρύους χειμώνες. Δεν νομίζω ότι η άνοιξη έχει καν έρθει σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Όλο αυτό σχετίζεται φυσικά και με όλο το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ε, εγκαίρως έρχεται, πολύ καλή στιγμή έρχεται η έκθεση αυτή και καλωσορίζω τις πτυχές της προστασίας του καταναλωτή και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε τις πρακτικές και να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να συνεισφέρει για να τονίσω τα όσα είπαν οι κύριοι Βαμπ και Στάιλερ. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην πτυχή του καταναλωτή, που είναι και η δικοτητά μας άλλωστε. Έχουμε πριν κάποιο καιρό εργαστεί επί της ενεργειακής χάρτας. Δεν ξέρω και τι έγινε με αυτό το έργο, μήπως ε, θα πρέπει να το διερευνήσει ο σύγητης. Αλλά πόσο θυμάμαι, τα κράτη-μέλη δεν ήταν πρόθυμα να έχουν ένα πρότυπο ευρωπαϊκό χάρτη και κατανοώ τους λόγους γι' αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε στην προηγούμενη θητεία μια κρόαση όπου είχαμε ομάδες ε, ε, ενεργειακών καταναλωτών και χρηστών που ήρθαν να μας μιλήσουν εδώ για, το θέμα της διαφάνειας, την αλλαγή, της αλλαγής παρόχου και για συνοριακά ζητήματα. Σίγουρα η ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είπε και η κυρία Στάιλερ, είναι ιδιαίτερα ενεργητική και επιδιώ και ασκεί δίωξη ε, κατά πολλών εταιριών ενέργειας και επιβάλλει και πρόστιμα όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν κακές ε, πρακτικές γιατί ε, υπάρχει διαφορά εκεί από το τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ε, όπου δεν είναι ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι καταρθώνουν ε, να πετύχουν μια καλή συμφωνία. Έτσι λοιπόν, αναλαμβάνω, αυτή την η ειδικότητά μας, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και επίσης σημείωσα στην έκθεση του κυρίου Κορέιντε Κάμπος το θέμα της αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών. Σε πολλές χώρες η εναλλακτική επίλυση διαφορών για τους καταναλωτές ενέργειας και η πρόσβαση σε αμερόληπτη παροχή συμβουλών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το της ενέργειας, πολύ περισσότερο από όλους τομές και για τις τηλεπικοινωνίες είναι σημαντική η διαφάνεια για τους καταναλωτές και ίσως και εκεί οι καταναλωτές να χρειάζονται ανεξάρτητες συμβουλές. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα άξιζε οι σκιώδεις και ο συγητής ίσως ε, να ε, τονίσουν το θέμα αυτό στη γνωμοδότηση και κυρίως το πώς σχετίζεται αυτό με την νομοθεσία για τους εναλλακτικούς μηχανισμούς διαφορών, για το EDR και ίσως θα πρέπει να είναι αυτό ένα τομέα όπου θα πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Σωστά τα είπε η κυρία Στάιλερ και για το κόστος της ενέργειας. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται το κόστος, αυτό είναι σαφέ. Και υπάρχουν καταναλωτέ που θέλουν να αγοράσουν πράσινη ενέργεια και ξέρουν, να ξέρουν ότι η ενέργεια που λαμβάνουν είναι πράσινη και τι πληρώνουν γι' αυτό. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολλά ζητήματα όπου το θέμα της διαφάνειας ε, και της ε, σήμανσης, της επισήμανσης δεν είναι ξεκάθαρα. Ίσως θα μπορούσε και ο συγητής να τα τονίσει αυτά, ιδιαίτερα εκ μέρους της Επιτροπής μας. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον από την Κομισιόν εδώ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Είστε εδώ για αυτό το θέμα για το επόμενο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει και να μας μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω μια απάντηση, μάλλον θα δώσω απαντήσεις, αλλά όχι απαραίτητα με τη σειρά που ακούστηκαν οι παρατηρήσεις, αλλά με τη σημασία των σημείων. Εγώ συμφωνώ με όσους πιστεύουν ότι η προτεραιότητα της γνωμοδότηση της δική μας πρέπει να είναι η ενίσχυση του συμφέροντος του καταναλωτή. Θα κάνω μία προσπάθεια για να ξαναβρω αυτόν τον ενεργειακό χάρτη του καταναλωτή. Θα πρέπει να κάνουμε και μία προσπάθεια να τονίσουμε την ελλακτική επίρρηση διαφορών και τις απαιτήσει διαφάνειας, που επίσης θα πρέπει να καλυπτούν και την πράσινη ενέργεια, καθώς όλες οι τεχνολογικές τροπές τελικά πληρώνονται από τον καταναλωτή αφενός και σε πολλές χώρες ε, αυτό ε, δημιουργεί το εξή αποτέλεσμα, ότι υπερβολικά πληρώνουν ο κάποιες από αυτές τις Δεν ε, είναι σαφή τα πράγματα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ, γιατί υπάρχει έλλειψη δαφάνειας σε όλα τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό συμφωνώ πως ε, αν είναι δυνατόν σε σχέση με την χρησιμοποίηση της πράσινης ενέργειας πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν μπορεί να χρησιμοποιεί πράσινη ενέργεια σε ψηλότερο κόστος ή αν πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί συμβατική ενέργεια σε χαμηλότερο κόστος. Γνωρίζοντα ε, βέβαια πόσο βλάπτει το περιβάλλον. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα επιλογής ε, του παρόχου, το switching. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μου έχουμε μια εμπειρία συλλογικής ελεγγύης, δηλαδή από τις 200.000 ε, οικογένειες που δημιούργησαν ομάδα για να μπορέσουν να οργανώσουν πιο πλέον μια συλλογική τέτοια αλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα αλλάξουν ε, πάροχο, αλλά θα έχουν περισσότερη πληροφόρηση και περισσότερο διαπραγματευτικό βάρος για να βρουν ένα πάροχο που θα τη συμφέρει καλύτερα ως προς το θέμα της ποιότητας τιμής. Και το κύριο εμπόδιο είναι το γραφειοκρατικό. Προσπάθησαν όλοι να βρουν μέτρα, να ε, ουσιαστικά αποθαρρύνουν τους καταναλωτές να αλλάξουν παρόχους. Και είναι απολύτως απαραίτητο εδώ η ρυθμιστική εξουσία του κράτους να ξεκαθαρίζει τις καταστάσεις αυτές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στο θέμα της ενεργειακή ανέχεια. Κύριε Σβάμπ, θα έχουμε πάρα πολύ καιρό για να μπούμε, μάλλον πολύ λίγο καιρό για το ποιο είναι το ο καλύτερος τρόπος να λύσουμε το θέμα της ενεργειακής ανέχειας. Θα έχουμε ανακοίνωση της Κομισιόν, περιμένουμε την ανακοίνωση αυτή και φυσικά θα ξεθάψουμε όλα τα επιχειρήματα υπέρ της οριζόντιας ή της ε, κάθετης μείωσης. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από ιδεολογική σκοπιά και είναι ιδεολογική η συζήτηση αυτή. Αν όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να μειώσουμε το υπερβολικό άχθος για τους ευπαθείς καταναλωτές, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως, την έχουμε μπροστά μας στη συζήτηση αυτή. Θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και τέλος, θα θέλω να υπενθυμίσω τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά στην ε, διέλευση της ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Ο κύριος Βάμπ υπενθύμησε ότι υπάρχουν κάποια κράτη προσπαθούν να θεσούν σε εφαρμογή μια πολιτική αυτάρκειας. Μια πολιτική ανεξαρτησία στον τομέα της ενέργειας για δύο λόγους. Είτε γιατί αισθάνονται καλά με την ε, σημερινή κατάσταση, είτε γιατί πιστεύουν ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στο μέλλον. Έτσι λοιπόν δημιουργώντας μια ανεξαρτησία, πιστεύουν ότι αισθάνονται καλύτερα. Δεν ε, μιλάω μόνο για τις ε, χώρες που μπήκαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις πιο παλιές χώρες, από τις πρώτες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν τη στάση αυτή. Είναι μια κοινή στάση, τη βλέπουμε σε όλα τα κρατη δεν μπορούμε να το κρύβουμε το πρόβλημα αυτό, αλλά αν η εσωτερική αγορά δεν έχει την ε, ικανότητα, αν δεν συγκεντρώνει τις επαρκείς δυνάμεις για να δημιουργήσει διασυνοριακά περάσματα και έχουμε γεωγραφικές συμφορήσεις και νομοθετικές συμφορήσεις, τότε εμείς ε, δεν θα καταφθάσουμε να δημιουργήσουμε μία κοινή αγορά ενέργειας και θα έχουμε πιο ακριβή ενέργεια τα επόμενα 30 χρόνια, το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε τον επαρκή τεχνολογικό ε, εξοπλισμό, είναι παροχημένος και πρέπει να τον ανανεώσουμε. Επομένως, είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί στο πώς ε, πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η εσωτερική αγορά ενέργειας, με ποια καθαρότητα πρέπει να δημιουργηθεί. Υπενθύμησε συνάδελφος ε, ότι υπάρχουν ε, διεθνή ε, ταμεία διεθνών ερευνητών που περιμένουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν μεγάλα ενεργειακά project και εγώ το πιστεύω αυτό εγώ νομίζω ότι το Connecting Europe με αυτά τα 9 δισεκατομμύρια που είχαν αρχικά προβλεφθεί είναι κάτι καλό. Θα είμαστε εμεί περίπου στα 5 δισεκατομμύρια, αλλά πρέπει να τα θεωρήσουμε ως seed money, ως αρχικά χρήματα χρηματοδότησης. Και θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση και από τον ιδιωτικό τομέα Εγώ σημείωσα όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης νομίζω ότι ήταν σημαντικό να τονίσουμε τις ενδυνάμει μελλοντικέ διαφορές, ε, δυσκολίες, με συγχωρείτε, που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε σε καλολημένα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 25 Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Good. thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας και τον εισηγητή αλλά και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους. 25 Απριλίου λοιπόν ε, υποβολή τροπολογιών, 29 Μαΐου θα ε, εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε. Στις 13 Μαΐου θα περνούσε από την Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποια συντονιστική δουλειά με τον εισηγητή και τους κοιόδης εκεί. Μπορεί να χρειαστεί λίγη δουλειά για να μπορέσουμε κάποιες από τις δικές μας απόψεις να τις περάσουμε, κυρίως για τα θέματα των καταναλωτών. Νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να προσθέσουμε κάτι στην ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Αυτά λοιπόν. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι μία νέα ε, έκθεση ε, πρωτοβουλίας ε, υπό την ηγεσία του Κορνέλη Ντε Ιόγκ, τον οποίο καλωσορίζω, για την προστασία των επιχειρήσεων κατά των παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Έχουμε κάποιο υλικό, μια σημαντική ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περσινή, ο κύριος Ντεγιόγκ θα την εξετάσει και εκείνη γιατί δεν έχουμε ακόμη απαντήσει σε αυτήν και ήταν μια σημαντική ανακοίνωση για την ε, εφαρμογή της εφιστάμενης νομοθεσίας κατά των παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στον εισηγητή, ποιος άλλος είναι εδώ από τους Κιώδης, ο κύριος Φαμπ, η κυρία Κόριν Λάγκεν που μιλά εκ μέρους του κυρίου Σφάμπ, ού είναι, είναι και εκείνη ε, ε, σκιώδη συγγήτρια. Εκ μέρους του κυρίου Σφάμπ, μάλιστα. Η κυρία Πρέντεκαστ δεν είναι εδώ. Η κυρία Πρέντεκας ε, νομίζω ε, αντικαταστάθηκε από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο σκιώδης και ο κύριος Μπίνεν είναι εδώ. είναι ένα πολύ αφοσιωμένο, είναι πολύ αφοσιωμένος συνάδελφος και βλέπω ότι είναι και πάλι εδώ. Ούτω ή άλλω θα συνεργαστούμε εμεί με τον κύριο Ντε για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για να μα πείτε ορισμένα πράγματα για τα βασικά στοιχεία που πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο συχνά υποτιμάται όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά γενικώ υποτιμάται. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Υπάρχουν απάτες, υπάρχουν καταγγελίες και στις κάτω χώρες. 3.000 καταγγελίες ε, λάβαμε ε, το 2008 Ήμασταν στις 11.000 το 2011 και 26.000 το 2012 μόνο κάτω χώρες λέω. Φέτος, 31 Μαρτίου, είχαμε ήδη φτάσει στις 8.000 καταγγελίες. Υπήρξε λοιπόν, ε, υπήρξαν καταγγελίες από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορες απάτες. Υπάρχει μια ε, προσπάθεια, μια απόπειρα που γίνεται όταν ένας ε, επιχειρηματίας ε, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα το οποίο τον ενημερώνει ότι αν θέλετε για παράδειγμα να ε, ολοκληρώσετε μία συνδρομή σας πρέπει να υπογράψετε αυτό το φάξ ε, και στο τέλος βλέπουμε ότι δεν είναι για τη σύναψη της σύμβασης αλλά για τη συνέχιση. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες που πέφτουν σε αυτή την παγίδα, δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο να ασχολούνται με αυτά τα θέματα, οπότε πολύ συχνά παγιδεύονται και αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. είναι μικρά τα ποσά, αλλά αν τα προσθέσει κανείς, 400 εκατομμύρια είναι οι απώλειες από τέτοιου είδους θέματα μόνο σε κάτω χώρες, λόγω τέτοιου είδους πρακτικών παραπλανητικών. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια αν προσθέσουμε τα ποσά απατών ε, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπήρξαν ήδη δύο ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν στο παρελθόν, το 2008, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και το ψήφισμα Μπουσούτιλ 2011 σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλεγε λοιπόν σαφοέστατα ότι ε, γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά ότι δεν υπήρχαν ε, ε, αρκετά βήματα που να έχουν γίνει. Ο κύριος Κάρας στο που είναι υπεύθυνος, που είναι πρόεδρος του Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έστειλε επιστολές στους διάφορους επιτρόπους προτείνοντας να ληφθούν κάποια μέτρα και το αποτέλεσμα ήταν η ανακοίνωση που πέρσι παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε κάποια ε, μέτρα να προτείνονται. Πιστεύουμε όμως ότι η έκθεση πρωτοβουλίας μας πρέπει να πάει λίγο πιο μακριά. Αυτό που απουσιάζει από την πρόταση της Επιτροπής είναι η πρόληψη. Προβλέπουμε εμείς κάτι στις ε, κάτω χώρες ε, για τους ε, επιχειρηματίες, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα γιατί προσβάλλει τη δυνατότητα του επιχειρήν των ανθρώπων αυτών. θα αρκούσε μέσω αυτής της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε δημιουργήσει για τους ε, επιχειρηματίες να είχαμε μία ε, τηλεφωνική γραμμή και για άλλους. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό πρέπει να συνοδεύονται αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές από βάσεις δεδομένων και πρακτικές που υπάρχουν για τα θέματα αυτά για να διευκολυνθούν τα, τα πράγματα για τους επιχειρηματίες ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα σύγκρισης. Αν κάποιος επιχειρηματίας λάβει ένα λογαριασμό που, τον οποίο δεν εμπιστεύεται πολύ, τουλάχιστον να μπορεί να πάει στη βάση δεδομένων και να συγκρίνει με άλλες περιπτώσεις. Όταν ε, παίρνει τηλέφωνο στην τηλεφωνική αυτή γραμμή, πρέπει καταρχάς να είναι δωρεάν το τηλεφώνημα. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, πρέπει να πάμε πιο πέρα από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωσή της. Η αστυνομία δεν ε, είναι πάρα πολύ πρόθυμη πάντοτε να καταγράφει τις ε, καταγγελίες ε, τέτοιου είδους επιχειρηματιών που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα μάλλον. Δεν είναι μία από τις προτεραιότητες για την αστυνομία. Υπάρχουν, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές να υπάρχει μια εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γνωρίζουν όλοι, να παραδεχθούν όλοι ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και ότι πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Χρειάζονται λοιπόν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις ε, υπηρεσίες καταστολής και δεν ισχύει κάτι τέτοιο στο πλαίσιο της ανακοίνωσης. Ο ρόλος της Ευρωπόλη είναι επίσης σημαντικός αλλά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν κάποια στοιχεία οργανωμένης εγκληματικότητας, υπάρχουν ε, συνέπειες επιβλαβή. πολλές. που χρήζουν προτεραιότητας. Και υπάρχει και το θέμα των ε, μεσολαβητών, των ενδιάμεσων με το ταχυδρομείο έρχονται τέτοιου είδους ε, επιστολές και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν παίζουν ρόλο ή συχνά έρχονται τεράστιες ποσότητες ε, ε, ε αλληλογραφίας που έρχονται από τους ίδιους ανθρώπους συνεχώς. μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για παράδειγμα. Υπάρχουν τρόποι. Ε, υπάρχουν τρόποι δράσης αυτών των εγκληματιών που μπορούν να αναγνωριστούν και σε επίπεδο πληρωμών αλλά και σε επίπεδο αλληλογραφίας. Εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε προτεραιότητες ε, που έχουμε λάβει από διάφορα δίκτυα και τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε, τις οποίες θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην ε, έκθεσή μας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, ομοιόμορφους κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως το πρόβλημα μπορεί να φτάσει ε, και μέχρι την Αυστραλία, γιατί ε, αυτά τα πράγματα δεν έχουν σύνορα ή σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτήν τη μορφή οργανωμένου εγκλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν το κάνει επαρκώς και το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είχα να πω. συνεχίζοντας αυτά που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα, μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας πει ποια θα ήταν ε, το, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της, ε, παρά, της ε, επέκταση στις οδηγίες του 2005 για τα ε, business to business, ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα. Νομίζω ότι δεν γίνεται ε, σωστή αξιολόγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι κάνει και τι δεν κάνει το κάθε κράτος μέλος. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Good. Μάλιστα. Έχουμε, καθώς φαίνεται, πολλά θέματα να επιλύσουμε με την έκθεση αυτή. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούσαμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκτενέστατη παρουσίασή σας. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Καταρχάς η κυρία Κόλιν Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Σβά που δεν μπορούσε να είναι εδώ που έπρεπε να φύγει. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τον ε, κύριο Ντεγιόν. Όντως χρειάζεται να δούμε τι γίνεται με τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Χρειάζεται εναρμόνιση, διότι η νομοθεσία να κράτος μέλος είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασία, ή διαφορετικά επίπεδα αντιμετώπιση από τις αρχές. Όσον αφορά τι διαβουλεύσει σε διασωνιαρικό επίπεδο, έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση των διασυνοριακών ε, περιπτώσεων και με αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως χρειάζεται να αλλάξει λοιπόν η νομοθεσία για την παραπλανητική διαφήμιση και αυτό πραγματικά το χαιρετίζουμε. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά. Καταρχάς μια νομοθετική πρόταση πρέπει να βασίζεται στην πλήρη εναρμόνιση με την νομοθεσία τη σχετική για τους καταναλωτές και τα καταναλωτικά προϊόντα και να τηρήσει την ε, νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να αποφευθούν οι αλληλοεπικαλύψεις. Έπειτα, υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας μαύρης λίστας επιχειρήσεων οι οποίες δρούν με παραπλανητικό τρόπο. Ένα, μια λίστα η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς και θα τονίζονται επίσης ε, σε τη διαστολή με αυτή και οι καλές πρακτικές. Τώρα όσον αφορά τον έλεγχο των επιχειρήσεων, εδώ σημασία έχει να αυξηθεί ο έλεγχος από τις αρχές, διότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τις ε, προϋποθέσεις και τους κανονισμούς που υπάρχουν. Επίσης, χρειάζεται ε, καλύτερη κωδικοποίηση, καλύτερη εξέταση, για παράδειγμα, της νομοθεσίας, η οποία θα ε, απορρέει και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ιδιαίτερα στον τομέα της συγκριτικής διαφήμισης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου ε, διαφημίσεις συγκρίνουν τις τιμές ανάμεσα σε διαφορετικούς απαρόχους υπηρεσιών. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει γραφειοκρατία και διοικητικός φόρτος. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα και μία λύση οικονομικά αποδοτική και σχετικά γρήγορη. Ο κύριος Φαμπ ευχαριστεί πάρα πολύ για την μέχρι τώρα εξαιρετική συνεργασία και προσβλέπει σε περαιτέρω συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας και εγώ να ευχαριστήσω και εκ μέρους εκείνου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο, ο κύριος Μάνιτό θα μιλήσει εκ μέρου του κύριου Ροσφόρ και ο κύριο Μπίλαν επίση. Η κυρία Στάιλερ, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε εκ μέρου τη κύρια Πέντεργκαστ. Κύριε Μπίλαν, έχετε το λόγο ω επίσημο σκιώδη συζητητή των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Και χαίρομαι πολύ που έχουν επισπευθεί οι εργασίες μας. Αναφέρομαι στην παρέμβασή μου για την γνωστή πρακτική των λάθος καταχωρήσεων σε Μητρώα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι απώλειες είναι εξαιρετικά υψηλές ε, και πολλές εταιρείε έχουν οδηγηθεί σε οικονομικά διέξοδα εξαιτία αυτής της λάθο ε, καταχώρηση. Στη γνωμοδότηση αυτή πιστεύω πως πρέπει να αναφερθούμε στα εξή σημεία. Πρέπει καταρχάς να λάβουμε υπόψη την ψηφιακή εσωτερική αγορά και τις καταχρήσεις που παρατηρούνται εκεί. Τις απάτες στον κυβερνοχώρο οι οποίες αυξάνονται. Έπειτα, η διασυνοριακή διάσταση του προβλήματος. Και εδώ αναφέρω την ανάγκη καλύτερης και στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα οδηγήσει στην καλύτερη καταπολέμηση της απάτης και της παραπλανητικής συμπεριφοράς στην αγορά και θα προστατεύσει τους καταναλωτές από τέτοιες πρακτικές και από πρακτικές που προέρχονται από τρίτες χώρες επίσης. Όσον αφορά τώρα την στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και την χρήση του συστήματος IMI, να πω ότι ως παλαιότερο εισηγητής στηρίζω την ιδέα αυτή απόλυτα. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά νομικά συστήματα Εν πάρει περιπτώσει όμως, σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες δεν χρησιμοποιούν μεσάζοντες, χρειάζεται να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές αποφεύγουν να προσφύγουν στο δικαστήριο λόγω του υψηλού κόστους μιας δίκης. αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. Επίσης, να στηρίξω την αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και να πω ότι προσβλέπω σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσουμε λοιπόν και τα, άλλη, και τα άλλα μέλη. Κυρία Στάιλερ, κύριος Μέντες. Κυρία Στάιλερ, έχετε το λόγο, αλλά πριν αρχίσετε να πω ότι καλωσορίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντάουν είναι εδώ πέρα από την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και, την υπεύθυ, και τον υπευθύνο τομέα, ο οποίος επίσης θα μας σχολιάσει τα όσα άκουσε. Κυρία Στάιλερ, όμως έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό, διότι για πολλούς από εμά, το θέμα μας αφορά άμεσα, έχουμε επηρεαστεί από αυτό. Ε, πριν από λίγες μέρες με προσέγγισε ένας ψηφοφόρος και μου είπε ότι η κατάσταση με τα Μητρώ έχει αλλάξει και ότι τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς μία γνήσια καταχώρηση από μία ψευδή και αυτό παρατηρείται και πραγματικά πρέπει να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, διότι λαμβάνουν επιστολές από, από δίθεν επιχειρήσεις που τους ζητούν διάφορα και θεωρούν πως είναι γνήσιες. Όμως αυτές δεν είναι και πραγματικά πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτές τις ε, ψευδείς επιστολές. Είναι απάτη αυτό, πρέπει να έχουμε καλύτερη οργάνωση, διότι πραγματικά υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτοί οι απαταιώνες, οι οποίοι καραδοκούν και εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης. Ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τους απαταιώνες που προσπαθούν να τους εκβιάσουν και να τους αποσπάσουν χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εγχείρημα αυτό και πραγματικά αν δείτε και τις περιπτώσεις στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες θα δείτε πόσο πολύ επηρεάζεται ο κόσμος από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάντος. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς έχω κάποιες άλλες υποχρεώσεις σήμερα, γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι συνέχεια παρόν. Όμως να πω ότι ο εισηγητής έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσίαση και θα ήταν καλό αν είχαμε και τη νομική υπηρεσία να εξετάσει τη νομική βάση της οδηγίας και ίσως να δούμε μήπως μπορούμε την οδηγία να την κάνουμε κανονισμό. Πιστεύω πως αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε και την ψηφιακή εσωτερική αγορά και θα ήταν πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εναρμονιστεί. Έπειτα, εφόσον εναρμονιστεί η νομοθεσία και είναι ίδια πανευρωπαϊκά, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσουμε αυτές τις απάτες. Και θα είναι Πιο εύκολο λοιπόν, αν είναι σαφέ, σαφής η νομοθεσία, θα είναι πιο εύκολη η ρύθμιση, πιο εύκολος ο έλεγχος και γι' αυτό θα μπορούσε ίσως να συσταθεί και ένας καινούριο οργανισμός. Για παράδειγμα, ένας ε, οργανισμός ε, όπου οι επιχειρήσεις θα ε, καταχωρούν πληροφορίες για περιπτώσεις απάτης ανακράτος μέλος. Και όταν κάποιος λαμβάνει απειλητικές επιστολές, για παράδειγμα, γιατί αν δεν πληρώσετε θα γίνει αυτό και εκείνο και θα γίνει προσφυγή και με... θα έρθει η πρακτική εταιρεία, τότε η επιχείρηση που πλήττεται από αυτό θα μπορεί να στέλνει αυτή την επιστολή σε μια κεντρική θέση όπου θα το αναλύει η ανάλογη ε, νομική υπηρεσία και θα αποφαίνεται εάν είναι ψευδή σε επιστολή, αν είναι γνήσια επιστολή και τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που είναι ψευδής. Αυτό θα αποτελεί ποινικό αδίκημα και θα κινείται ποινική διαδικασία. Αυτό θα μπορούσαμε λοιπόν να το συνοψίσουμε όλο σε κανόνες. Ωραία. Νομίζω ότι Ακούσαμε πολλές απόψεις και αυτό που είπε ο κύριος Μάντερ στο τέλος. Αυτό σχετίζεται με κάποια θέματα αλλά ότι προσπαθούν κάποιοι ε, να θέσουν διασυνοριακά σε εφαρμογή την εκτέλεση δραστικών αποφάσεων. Υπάρχουν και κάποια νομικά θέματα που πρέπει να σκεφτούμε για το γεγονό ότι μικρέ ε, επιχειρήσει δεν είναι σε θέση να υπερασπίσουν τον εαυτό του σε μια δικαιοδοσία. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά τελικά υποχωρούν, εκφοβίζονται από αυτά τα αιτήματα πληρωμών και όταν ε, μιλάμε για αυτές τις απάτες καταλόγων, ε, Αρκετέ κυβερνήσει, όπω η Ολλανδική, η Ισπανική έχουν αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και τελικά έδωσαν συμβουλέ ε, στι μικρέ επιχειρήσει να μην το πληρώνουν και να στέλνουν μια επιστολή όπου θα αρνούνται την πληρωμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αποτελεσματική διαδικασία ανάκτηση, αλλά με ενδιαφέρε θα με ενδιαφέρει αυτό να το δούμε, αλλά υπάρχουν πολύ πλοκανομικά θέματα και θα πρέπει ίσως ε, να καλέσουμε και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, να τα εξετάσουν αυτά. Μόλις έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα και πρόσεξα ότι αναφερθήκατε και στο θέμα της ε, επιβολής χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Europol και τις αστυνομικές αρχές. Ίσως λοιπόν, Ντένις, θα πρέπει να κάνεις και κάποια καμπάνια στις άλλες επιτροπές για να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η συνολική εντύπωση που δίνεται είναι ότι οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις είναι μια ομάδα που συχνά παραμελείται σε αυτές τις δραστηριότητες. Και Ξέρουμε ότι αυτές οι απάτες ε, καταλόγων ε, είναι πολύ συγκεκριμένος κίνδυνος, αλλά υπάρχουν και άλλου είδους απάτες. Ένας άλλος ε, τομέας που ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και το θέτω επιτάπητος, για να υπενθυμίσω σε όλους ότι όταν είχαμε το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και τις καθολικές υπηρεσίες, είχαμε εκεί μια διάταξη διευκόλυνσης όπου τα κράτη-μέλη οι ρυθμιστικές αρχές ε, των κρατών μελών θα μπορούσαν ε, κάποια από τα μέτρα προστασίας για τις τηλεπικοινωνίες ε, να τα επεκτείνουν για να καλύψουν και τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προχωρήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια πόσες αρχές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία. Και ίσως θα μπορούσαμε να γράψουμε στην κυρία Κρούς και να μάθουμε γιατί αυτό το έχει ζητήσει αυτή η Επιτροπή Καθώ οι τηλεπικοινωνίες, αλλά στο μέσο που νομίζω ότι μικρές επιχειρήσεις ε, μπορεί να είναι θύμα ε, τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών στη διαφήμιση. Έχουμε λοιπόν μια σωρία θεμάτων, αλλά νομίζω ότι το τελικό πρόβλημα είναι πως ε, χρηματοδοτούμε πρόσθετε δραστηριότητες προστασίας για τις μικρές επιχειρήσεις τη στιγμή που έχουμε περιορισμό στους πόρους μας. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για την αποπτία της αγοράς. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ διστακτικά να επενδύσουν παραπάνω σε αυτούς τους τομείς. Θα πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες σκέψεις και από μένα. Τώρα με χαρά να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Να σας δώσω την ευκαιρία να σχολιάσετε. Για όσοι υπόθηκαν μέχρι τώρα και κατόπιν θα ξαναδώσω το λόγο στον συγητή, στον κύριο Ντεγιόν για το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ, κύριε Ντόνι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Καταρχήν, η Κομισιόν πιστεύει ότι πράγματι στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών και εκατοντάδες μικρέ επιχειρήσεις είναι θύμα τέτοιων πρακτικών καθώς έχουν ε, διευρυνθεί οι μαζικές πρακτικές, έχουμε φτάσει στον αριθμό των 6 εκατομμυρίων ετυπών ε, ετησίως ε, και τέτοιε μικρέ εταιρείε μπορεί να χρειάζεται να πληρώνουν από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ και είναι πολύ τεράστιο το ποσό για τι μικρέ επιχειρήσει. Επίση, είχαμε 30.000 καταγγελίε. Έγινε μία μελέτη Από την πλευρά της Κομισιόν το 2011 ξεκινήσαμε δημόσια διαβούλευση και εκεί το 81% όσων απάντησαν θεώρησαν ότι το πρόβλημα ε, των παραπλανητικών πρακτικών είναι σημαντικό και το 79% ζήτησαν δυνάμωση της προστασίας των ε, μικρών επιχειρήσεων. Γι' αυτό, σύμφωνα με τη δεσμευσή μας, δικαιοσύνη για την ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι πρέπει η πολιτική μας να συνδυάσει την προστασία των καταναλωτών με την προστασία των πολιτικών. Στην ανακοίνωση που παρουσιάσαμε, δεχτήκαμε ότι σήμερα το μόνο νομοθέτημα που υπάρχει σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει τι επιχειρήσει από τι παραπληκτικέ πρακτικέ ε, marketing είναι η οδηγία για την ε, συγκριτική διαφήμιση και είναι ένα θέμα που δίνει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασία. Όμω, ε, το λέμε ανοιχτά, γνωρίζουμε του περιορισμούς τη οδηγία αυτή αφενός ε, κάποιοι κανόνες από αυτή την οδηγία μπορεί να μην είναι αρκετά ξεκάθαρη και από την άλλη, η εφαρμογή σε διασυνορικό επίπεδο έχει δείξει ότι υπάρχουν παραθυράκια. Δεν υπάρχει νομική βάση για τα κράτη-μέλη, για τι αρχέ των κρατών μελών να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίση, υπάρχει απουσία σύγκληση ε, των μοντέλων επιβολή στα κράτη-μέλη και γι' αυτό Πέρσι τον Νοέμβριο δημοσίευσα μια ανακοίνωση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Στην ανακοίνωση τονίζονται δύο κύριε προτεραιότητες. Καταρχήν, θα θέλαμε να εξετάσουμε το θέμα της επιβολής τη εκτέλεση πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ισχύουν οι κανόνες ε, και ότι δεν μπορούν να κρυφτούν οι παραβάτες πίσω από τα σύνορα, θέλουμε να δώσουμε στις αρχές των κρατών μελών ένα πιο διορθωτικό πλαίσιο και μια νομική βάση για να συνεργαστούν αλλά και εξουσίες για να σταματήσουν αυτές τις παραπλανητικές πρακτικές. Δεύτερον, θέλουμε να δούμε το ουσιαστικό τμήμα της νομοθεσίας και πιστεύουμε ότι προκειμένου να αυξήσουμε την ασφάλεια δικαίου, πρέπει να καλύψουμε τα φυστάμενα κενά για να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες, ε, ίσως ε, απαγορεύοντας με τη μορφή και μιας μαύρης λίστας μια σειρά παραπλανητικών πρακτικών. Και τέλος, εξετάζουμε και τις ποινές για να διασφαλίσουμε ότι είναι αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές. Αυτό είναι το πλαίσιο των δύο προτεραιοτήτων Όμω, λεχθέν των αυτών, καλωσορίζω τα σχόλια του εισηγητή, βεβαίως και εξετάζουμε το θέμα της πρόληψης, της πολιτικής και είμαστε σε επαφή με το κέντρο στην Ολλανδία για την πρόληψη της απάτης. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε ότι οι πιο επιτυχείς προληπτικές δράσεις ελήφθησαν από τις ίδιες τις οργανώσεις των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι οι οντότητες ε, που είναι πιο κοντά στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις έχουν τα πιο κατάλληλα εργαλεία για να σχεδιάσουν αυτά τα προληπτικά μέτρα, όπως είναι οι hotlines. Γραμμής εκτακτής ανάγκης. επίση, εξετάζουμε το θέμα της διεθνού συνεργασίας, αναπτύσσουμε αυτή την πολιτική. Επίσης, ε, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή να λαμβάνει δράση κατά αυτό των πρακτικών και αναζητούμε τους διάβλους ε, για επικοινωνία και συνεργασία με ΙΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία για τη συνεργασία με τη Europol. Και αυτό θα είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε για να αντιμετωπίσουμε το ποινικό σκέλος του προβλήματος και φυσικά ε, το ζήτημα του δικαίου για το μάρκετινγκ πρέπει να συμβαδίσει και με το ποινική πτυχή. Σε ό,τι αφορά την οδηγία περί των εμπορικών πρακτικών. Να επιστήσω την προσοχή σας, η Κομισιόν μόλις δημοσίευσε την ανακοίνωση και την έκθεση για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και εκεί υπογραμμίζουμε το πώς κατανοούμε την εφαρμογή της οδηγίας που λέει ότι πιστεύουμε ότι οι σημερινοί κανόνες φαίνεται να είναι αποτελεσματικοί αλλά υπάρχει πρόβλημα επιβολής και επίσης και στο ρόλο της Κομισιόν για την επιβολή και προσπαθούμε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε αυτή την επιβολή του νόμου και να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά με τα κράτη-μέλη. Βεβαίω και καλωσορίζω τα σχόλια σε ό,τι αφορά την ψηφιακή αγορά. Αν ε, έχουμε μία διαίρεση των κανόνων για το B2B, θα πρέπει να εξετάσουμε και το online marketing, το επιγραμμικό marketing. Επίσης, ε, δεχόμαστε, παραδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό όταν ε, προετοιμάσαμε τα μέτρα επιβολής ε, και το, τους πιθανούς τρόπους συνεργασίας από το τομέα, θέλαμε να έχουμε ένα όσο δυνατόν πιο ελαφρύ σύστημα, αλλά και στο δυνατόν πιο αποτελεσματικό, δηλαδή να μην θέσουμε υπερβολικό άχθος της δικής των κρατών μελών που έχουν ελπίσει πόρους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ περιεκτική σας απάντηση και γιατί μας είπατε και ποια είναι η θέση σας ε, για διάφορα θέματα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, νομίζω όχι. Αν θυμάμαι, μας υποσχέθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπή και στην ανακοίνωση αυτή ότι θα υπήρξε, θα υπήρχε νομοθετική πρόταση πριν από το 2013 ακόμα εξακολουθεί να αποτελεί φιλοδοξία σε αυτό. Ναι, η φιλοδοξία μας είναι... Αυτή τη στιγμή είμαστε στη μελέτη αξιολόγησης και αν ε, αυτή επιβεβαιώσει την ανάγκη για νομοθετική δράση, ναι, το πρόγραμμά μας είναι να υποβάλουμε πρόταση φέτος. Οπότε αν εγκριθεί η γνωμοδότηση του κυρίου Ντε θα συνεισφέρει στη διαδικασία, να μην χάνουμε το χρόνο μας δηλαδή. Ναι, πράγματι, λέει ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μάντερς, συγγνώμη, δεν άκουσα απάντηση στο ερώτημά μου για τον ε, κανονισμό. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε στον κύριο Μάντες. Πάντοτε κάνει αυτή την ερώτηση. Οπότε όποιο έρχεται εδώ από την Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει. Μήπω μπορείτε να την επαναλάβετε. Να το κάνω, ναι. Είπα απλώ ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς που δεν έχει σύνορα πρέπει να εισαγάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο εναρμονισμένη νομοθεσία και ίσως καλύτερα να το κάνουμε μέσω κανονισμού αντί για ε, οδηγίας. Ε, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τη νομική βάση για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ερώτησή Με Ευχαριστώ πολύ, λέει ο εκπρόσωπος Επιτροπής, για την αλλαγή από κανονισμό σε οδηγία. Πρέπει να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα εθνικής νομοθεσίας που καλύπτει όχι μόνο τον τομέα αυτό, αλλά την ευρύτερη έννοια του ε, θεμητού ανταγωνισμού που καλύπτει κάποιες πρακτικές εκτός ε, του μάρκετινγκ. Και δεν θα θέλαμε να επηρεάσουμε το σύστημα αυτό, το οποίο είναι αρκετά περιεκτικό και αποτελεσματικό. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η δράση στον τομέα των ε, παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ θα έπρεπε κάπως να συμπληρώνει τους ε, υπάρχοντες κανόνες. Λόγω αυτού πιστεύουμε ότι κατά την, για, την ώρα ε, το καλύτερο μέσο είναι η οδηγία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί η απάντηση αυτή του κυρίου Μάντες, αλλά, το κύριο Μάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε. Κύριε Ντε μήπως μπορείς να μας συνοψίσεις και να μας πεις ε, για το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Ευχαριστώ Μάλκολ. Ευχαριστώ και όλους όσους πήραν το λόγο. Νομίζω ότι υπήρξαν ε, διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές προτάσεις. Δυστυχώς ε, υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορώ να χρησιμοποιήσω στο, στην έκθεση πρωτοβουλίας και κάπως με περιορίζει αυτό. Όσον αφορά τώρα τις λεπτομέρειες ε, της πρότασης της Επιτροπής, ναι, δεν μίλησα πολύ, είπα ότι θα έπρεπε να πάμε πολύ πέρα από αυτό, αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ χρήσιμα αυτά που έχει συμπεριλάβει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Εγώ έχω πάντοτε την τάση να είμαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τις δαπάνες. Δεν πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες ε, δαπάνες. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε απώλειες 400 ε, ε, εκατομμυρίων μόνο για μια χώρα όπως οι κάτω χώρες, καταλαβαίνετε ότι το, το, το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου έκανε εντύπωση που μας ζητήθηκε και μας να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και η Λίμπε μπορεί να ενδιαφερόταν και εκείνη. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Γραμματεία, το σχέδιο γνωμοδότησής μου δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου θα σας το παρουσιάσω, θα μεταφραστεί. 29 και 30 Μαΐου θα σας παρουσιαστεί αν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές, πρέπει βέβαια να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα γιατί υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. Αν σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε στο, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε παραπάνω, ακόμη και αν ε, η πρόταση της Επιτροπής γίνει στο πλαίσιο του 2013. Καλό είναι να έχουμε και την άποψη των υπολείπων επιτροπών, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τις εργασίες μας άλλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, να έχετε υπόψη ότι ενδεχομένω να έχουμε μια νομική πρόταση μέχρι τότε. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε λοιπόν. Και να δούμε και το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις ε, δικές σας ε, τροπολογίες και την εξέτασή τους και το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ όμως, όπως και να έχει, που ανοίξατε αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ σημαντικό και καινοτόμο θέμα για την Επιτροπή αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν με δύο θέματα που συνδέονται για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας εντός της ώρας. Έχουμε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την οδηγία και την γνωμοδότηση για αυτή, που, ε, η γνωμοδότηση η οποία έχει γίνει για την ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Υπάρχουν όλοι οι συγητές, οι σκιώδει συγητές, ο κύριο Κάρα είναι από το ΕΛΚ. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλου ενεργού σκιώδει Θα σα δώσω το λόγο αμέσω Έχουμε επίση και τη γνωμοδότηση για τα έγγραφα με βασικέ πληροφορίε σχετικά με επενδυτικά προϊόντα. Ξέρω πω ο κύριο Παντζέρη λείπει. Ο κύριο Κονφεράτη όμω θα μιλήσει εκ μέρου του ω εισηγητή. Ξέρω πω η κυρία Πιτικάινεν είχε άλλη επιτροπή σήμερα, αλλά πιστεύω πω η κυρία Λάγκεν θα μιλήσει εκ μέρου τη. Ο κύριο Μπουζόη επίση λείπει. Δεν ξέρω ποιο θα μιλήσει για του φιλελεύθερου. Αυτό που προτείνω είναι να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε τροπολογίες να συζητήσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν κυρία Στάιλερ, κύριο Κάρας και μετά οτιδήποτε άλλο έχουμε να πούμε για τις εμβαστικές τροπολογίες και μετά θα δούμε και τη γνωμοδότηση του κυρίου Παντζέρη. Επίσης έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, νομίζω ο κύριος Βανχούλα ή όχι. Όχι, ο κύριος Βανχούλα πήρε σύνταξη. Μάλιστα. Ποιος θα μιλήσει λοιπόν. Μου Steve Ryan, Steve Ryan. Θα καλύψετε λοιπόν και τα δύο θέματα. Ή όχι. Ποιος θα κάνει το θέμα για τις ασφάλειες. Ο συνάδελφος. Πολύ ωραία. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση λοιπόν. Κυρία Στάιλερ, έχετε το λόγο και μετά ο κύριος Κάρας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους σκιώδεις εισηγητές. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μαζί συμβαστικές τροπολογίες και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κάρας εδώ που ήταν παρόν σε όλες τις ε, συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών. Ξέρω πόσο ε, φορτωμένο είναι το πρόγραμμα όλων σας. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα το κείμενό σε συμβαστικέ ε, τροπολογίε και αυτό εν μέρει επειδή ορισμένοι εισηγητέ δεν ήταν τόσο ενεργοί όσο ο κύριο Κάρα και δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω όμω ότι μέχρι τις 25 Απριλίου που θα γίνει και η ψηφοφορία να μπορέσουμε να έχουμε το τελικό κείμενο. Ξέρω ότι υπάρχει σύγχυση με ορισμένε συμβαστικέ τροπολογίε και θα προσπαθήσω να δω αυτές που θεωρώ σημαντικότερες. Για παράδειγμα, συμβαστική τροπολογία 1 για τα συγκριτι... τους συγκριτικούς ιστότοπους. Τη θεωρώ πολύ σημαντική. Έχουμε βάλει μια επεξήγηση για τις πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα και ότι τα ιστότοποι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται ως ε, μεσολαβητές αλλά πρέπει να φροντίσουμε να συμπεριληφθεί ο εμπορικό χαρακτήρας τους. Επίσης, μετά συμβαστική τροπολογία 2 για, την προσωπική, για τις προσωπικές συμβουλές, υπάρχει ο ορισμός ο οποίος μας δημιούργησε πρόβλημα, ο ορισμός του συμβιβασμού. Επίσης, για το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις πρακτικές, φυσικά καθώς κοιτούμε το τι γίνεται με τη σύνδεση και την ομαδοποίηση. Έχουμε προσπαθήσει και εκεί να συμβιβαστούμε στο θέμα της σύνδεσης, διότι όταν αγοράζεις ένα προϊόν το οποίο είναι συνδεδεμένο με κάποιο άλλο, το πρόβλημα που προκύπτει για την προστασία των καταναλωτών είναι οι επιλογές που αυτοί έχουν. Και παρότι προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε σε αυτό το ζήτημα και να το αντιμετωπίσουμε, τα συνδεδεμένα προϊόντα δηλαδή, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν την επιλογή όταν αγοράζουν ένα προϊόν που είναι συνδεδεμένο με κάποιο άλλο να μην πάρουν και τα δύο, αν δεν το επιθυμούν. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του ανταγωνισμού το οποίο αντιμετωπίζεται σε αυτήν την τροπολογία. Επίσης έχουμε 16 συμβαστικές τροπολογίες να σας πω συνολικά. Οι 7 είναι δεν χρειάζεται εξήγηση. Ενσωματώνεται λοιπόν στην ε, ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Τώρα στο άρθρο 7, η τροπολογία του άρθρου 7 μας ε, δημιουργεί κάποια σύγχυση για την, ε, που αφορά την παράγραφο 1F και θα σας τα πει και ο κύριος Κάρας με τις απολαβές είναι το θέμα. Εδώ προσπαθήσαμε να την αναδιατυπώσουμε και να αναφερθεί ότι να αναφερθεί ρητά η αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αίτημα του ενδιαφερόμενου, του καταναλωτή δηλαδή. Όμω ε, πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια σύγχυση, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε πρώτου προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα για αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία. Τώρα, τροπολογία 9 να το κοιτάξουμε και αυτό. Πιστεύω επίσης πως ε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Έχουμε αλλάξει κάποιες λέξεις, οι οποίες ήταν λίγο προβληματικές. Ορισμένοι είχαν ευαισθησία απέναντι σε αυτές. Μετά, κάτι που μας έχει μπερδέψει είναι τα ζητήματα με τους ε, μεσάζοντες τους διοικητικού διακανονισμούς και την προσπάθεια για εκτόνωση των διαφορών. Μετά 15 και 16 είναι απλό σχετικά το θέμα, μιλά για τις απολαβές. Αυτό που προσπαθήσαμε εδώ να κάνουμε και βασίζεται στο άρθρο 17 ήταν να δώσουμε σαφήνεια. Καταρχάς, να, υπάρχουν απο, ε, να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις απολαβές για προϊόντα ζωής και όχι. Φυσικά για τα προϊόντα, που αφο, για τα προϊόντα ζωής ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στις απολαβές. Για τα υπόλοιπα προϊόντα έπρεπε να βρούμε κάποιο συμβιβασμό όσον αφορά τις απολαβές και αυτό φαίνεται και στο άρθρο 17 και απορρέα από αυτό. Γενικά στο συμβιβασμό που προσπαθήσαμε να έλθουμε, θεωρώ σημαντικό το ότι το καταφέραμε στα πιο αμφιλεγόμενα σημεία και έχουμε καταφέρει να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι αυτό που προσπαθούμε εν τέλει να κάνουμε είναι να δούμε τους καταναλωτές και πώς θα προστατεύονται οι καταναλωτές από όλα αυτά τα διαφορετικά προβλήματα. Έχουν ξεσπάσει σκάνδαλα τα οποία έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ασφαλιστικά προϊόντα και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτό. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη του κυρίου Κάρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ότ Μαρκάρας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, συνάδελφοι και συγγήτρια. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία και για την ετοιμότητα που είχατε για συνεργασία και τα ανοιχτά σας αυτιά. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα μας, βρισκόμαστε φυσικά σε περίοδο κρίσης και είναι απαραίτητο να ξαναχτίσουμε την πίστη των καταναλωτών στα ασφαλιστικά προϊόντα και στην ασφαλιστική αγορά. Αυτό είναι ένας από τους ε, κυρίους στόχους μας. Η επεξεργασία της ε, οδηγίας, λοιπόν, για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μιλήσατε ήδη για τις ε, συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Το μόνο που μένει είναι να τις ολοκληρώσουμε. Ορισμένα θέματα συγκεκριμένα που αναφέρονται σε άρθρα λείπουν, ε, μας μένουν ακόμα να ολοκληρώσουμε. Για παράδειγμα την τιμολόγηση. Επίσης, το πεδίο εφαρμογής δεν συμπεριλαμβάνονται οι σύνδεσμοι καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται μέχρι τώρα. Μετά, ορισμός των ε, προϊόντων, των συνδεμένων προϊόντων έχει γίνει πιο αυστηρός, πιο συγκεκριμένος και είναι πιο, αυστηρές, πιο αυστηρά τα, τα κριτήρια τα οποία θα επιτρέπουν τη σύνδεση ενός ασφαλιστικού προϊόντος με ένα άλλο. Επίσης, η σχέση των ασφαλιστικών προϊόντων με τους καταναλωτές πρέπει να συνάδει με την οδηγία. Αυτό θα το ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Αλλά να πω ότι χρειάζεται προσαρμογή καταρχάς με την ε, νομοθεσία και από την για να αποφευχθεί και περισσότερη γραφειοκρατία και ε, αλληλοεπικαλύψεις. Όσον αφορά τις ε, πρακτικές, μας ενημέρωσε η συγγήτρια, εμείς ζητούμε την ενημέρωση ε, κατόπιν αιτήματος. Μετά για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. και αυτές πρέπει να γίνουν. Όμως πρέπει να προσέξουμε, με ορισμένες, ε, να προσέξουμε ορισμένους τομείς οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με αυτά που προτείνουμε. Τώρα όσον αφορά τις, ε, την ασφαλιστική μεσητεία. η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων έχει ασχοληθεί με το θέμα και μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ε, καταλήξει στην ε, πρόταση για διαγραφή του σχετικού σημείου διότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, Γιούρι δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογής ήταν ιδιαίτερα μεγάλο όσον αφορά την ασφαλιστική μεσητεία και αυτό ενδεχομένως προκαλέσει άνισες συνθήκες ανταγωνισμού και μείωση της διαφάνειας για τα εν λόγω προϊόντα. Και αυτό ενδεχομένως ε, λειτουργήσει και, ε, οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών. Επίσης, πληρωμές είναι ένα θέμα για το οποίο συμφωνούμε με την ε, Επιτροπή Γιούρη. Γενικά πάντως να πω ότι έχουμε επεξεργαστεί το θέμα αρκετά και πιστεύω πως ε, η Επιτροπή Γιούρι έχει κάνει και αυτή πολύ καλή δουλειά. Συμφωνούμε και εμείς μαζί της και ε, πραγματικά υπομονούμε να ολοκληρωθεί το πακέτο. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητές και τον συνάδελφο Κάρας. Ξέρω πως ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό, διότι είναι και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομικών, και Υποσχέσεων και ξέρει πολύ καλά τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που εξετάζουμε τώρα. Θα είμαι σύντομος, θα κάνω μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, ο συμβιβασμό σχετικά με την καταχώρηση σε μητρώα των διαμεσολαβητών ναι, πρέπει να γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία. Εγώ ε, υποστηρίζω απόλυτα αυτό που έχει προταθεί τώρα όσον αφορά την επίλυση των διαφορών. Εδώ έχω κάποιες ε, αμφιβολίες, διότι στην οδηγία αναφέρονται οι διαφορές ανάμεσα σε καταναλωτές. Και εδώ πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε αναλόγως το κείμενο. Ε, κατά τα άλλα συμφωνώ με τον κύριο Κάρας για αυτά που έχει προτείνει τώρα. Όσον αφορά τι επιχειρήσης προ καταναλωτέ. Ένας πελάτης μπορεί να είναι και μια επιχείρηση και ένα καταναλωτή απλώς καταναλωτής. Γι' αυτό πραγματικά εδώ σας καλώ να προσανατολιστούμε στο κείμενο της οδηγίας και να βάλουμε τον καταναλωτή στο επίκεντρο. Έπειτα, όσον αφορά την πληροφόρηση του καταναλωτή, εγώ πιστεύω ότι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ε, με άλλα λόγια, πρέπει να έχει το δικαίωμα να υποβάλει να υποβάλει ερώτηση και να λαμβάνει σαφείς και ξεκάθαρε απαντήσεις όσον αφορά το κόστος και τις λεπτομέρειε των προϊόντων που έχει αγοράσει. Τώρα για την διαγραφή του άρθρου, της παραγράφου 1 1D του άρθρου 1 για τα μη ε, για τα προϊόντα, για τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν αφορούν ε, ασφάλειες ζωής και εδώ πρέπει να προσέξουμε να δούμε τις ε, λεπτομέρειες. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Ρόιτσεβα. Ευχαριστώ. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο των συγκεκριτών στον τομέα αυτό. Αλλά θέλω κάτι να τονίσω, το οποίο επανέρχεται ως μπούμεραγκ. Η... Είπε ο γερμανό συνάδελφο ότι ο καταναλωτή μπορεί να είναι και πελάτη. και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρε όπω η Γερμανία. Το καταναλωτικό δίκαιο συμπεριλαμβάνει και τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει, αλλά σε άλλε χώρε εξαρτάται ε, από το δικαιό του αν θα τι συμπεριλάβουν ή όχι στην τσεχική δημοκρατία. Δυστυχώ δεν έχει γίνει δυνατό ακόμη να ισχύσει κάτι τέτοιο. Αν δεν εναρμονίσουμε λοιπόν τον ορισμό και το ποιε οντότητε εμπίπτουν στο καταναλωτικό δίκαιο, δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ούτε επί άλλων μέτρων. Εδώ θα λοιπόν, θέλω να ρωτήσω του συναδέλφου, να ζητήσω μάλλον από του συναδέλφου να είναι ευέλικτοι, γιατί είναι ένα είδο κοκκίνη γραμμή. Εμεί προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα να σκεφτούμε λοιπόν έναν ορισμένο ορισμό των οντοτήτων που εμπίπτουν στο καταναλωτικό δίκαιο. Βέβαια, εγώ προτείνω να ανήκουν εκεί οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ε, γιατί ε, τελικά οι καταναλωτές είναι ηριγμένοι όταν ε, μπαίνουν σε διενέξεις, όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορές με επιχειρήσεις που έχουν, ξέρετε, πολύ ισχυρούς δικηγόρους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για αυτές τις λεπτομέρειες. Και ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο από μένα. Στις συμβαστικέ τροπολογίες τη ε, κυρίας Τέλερ, στην υπερφών 2, μιλά για την ε, σύσταση που δίνεται σε έναν πελάτη, αλλά κατόπιν έχουμε και έναν ε, ορισμό για την προσωπική συμβουλή και φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση μεταξύ των δύο και θα ήθελα να μου πει τι ακριβώς είχε εδώ κατά νου ως προς τους ορισμούς ε, γιατί το θέμα αυτό της ε, της συμβουλών είναι ζωτική σημασία για όλη τη δουλειά που κάνουμε για τους καταναλωτές και για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για τη σημασία του να παρέχουμε στους ανθρώπους τις κατάλληλες ε, συμβουλές και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ανεξάρτητη συμβουλή και τη μεροληπτική συμβουλή. Επίσης, επομένως, δεν ήμουν σίγουρος τι γίνεται ακριβώ με του ορισμού και τι αντικαθιστά τι. Ίσως να θέλετε να το σχολιάσετε αργότερα. Τώρα, και ε, θα ε, καλούσε ίσω και τον κύριο Ρέα να κάνει κάποια σχόλια, αν συμφωνείτε κύριε Τάιλερ, και κατόπιν θα σα δώσω το λόγο για να συνοψίσετε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κύριε Ράιν. Ευχαριστώ. Να πω από την αρχή ότι αυτό αποτελεί ένα τμήμα δέσμες μέτρων όχι μόνο με την πρόταση που συζητάμε σήμερα για την περίπτωση, αλλά και για την πρόταση MIFID, που είναι ένα κυρίως στοιχείο του πακέτου. Και σε ορισμένα σημεία πρέπει να κάνουμε κάποιο παραλληλισμό σε σχέση με το τι θα προτίσουμε για την πρόταση AMD και για τη ΜΥΦΙΔ. Φυσικά αυτή είναι μια πρόταση που σκοπεύει στην προστασία των καταναλωτών και στην αυξανόμενη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Κάποιες τροπολογίες στοχεύουν περισσότερο στην προστασία των καταναλωτών, ενώ άλλες επιδιώκουν να μειώσουν το άχθος στις επιχειρήσεις, κυρίως στις ΜΜΕ. Δεν θα σας εκπλήξει να ακούσετε ότι η Κομισιόν ε, περισσότερο ότι είναι προς την προστασία των καταναλωτών, γιατί φυσικά όταν παρουσιάσαμε την πρότασή μας, ε, παρουσιάσαμε και μία πλήρη μελέτη αντικτύπου που αξιολόγησε καθολικά τον αντίκτυπο, εξαντλητικά τον αντίκτυπο στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει και θεωρούμε ότι η πρόταση τη Κομισιόν πετυχαίνει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυξημένη προστασία των καταναλωτών και του άχθου στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Όπω λέγεται στη μελέτη δικτύπου για κάποια συγκεκριμένα τώρα σημεία. Οι κύριες πτυχές της πρότασης της Κομισιόν είναι καταρχήν η επέκταση του πεδίου εφαρμογή σε σχέση με την φυστάμενη MD για να καλυφθούν όλοι οι διαβλοί πωλήσεων, των ασφαλίσεων αλλά και η επικουρική υπάροχη παροχή ασφαλίσεων, όπως είναι ε, κάποια γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων ε, ή τα ταξιδιωτικά γραφεία. Δεύτερο στοιχείο της πρότασης της Κομισιόν είναι η τα ταξιδιωτικα γραφεια δευτερο στοιχειο της πρωτης διαφάνεια και σχετικά με την αποζημίωση και τις προμήθειες. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία θα είχαμε ένα ερωτηματικό στο νου μας σχετικά με την προστιθέμενη αξία της πρότασης. Σε σχέση λοιπόν με τη διαφάνεια των αποζημιώσεων, των αμοιβών, Πιστεύουμε ότι μετά από επαρκής ε, περίοδους μετάβασης για, τι για τις ασφάλειες, ε, εκτός από τις ασφάλειες ζωής, ε, θα πρέπει να έχουμε επαρκή διαφάνεια για τις αμοιβέ χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής ε, να το ζητήσει αυτό, να υποβάλει αίτημα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ίσους κανόνες για όλους μεταξύ των διαφορών διάβλων πωλήσεων και πλήρη εξουσία στον καταναλωτή για να έχει μια κατάλληλη συμφωνία με τον πολίτη ανεξάρτητα από το είδος του πολίτη. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το κόστος, η πλήρη τιμή του προϊόντος, να ξέρει ποιο είναι το περιθώριο του κέρδους ε, μέσα στο προϊόν. Αυτό είναι λοιπόν στην καρδιά της πρότασης της Κομισιόν. Αν το αφαιρέσετε αυτό ή αν αποδυναμωθεί αυτό, θεωρούμε ότι είναι κέριο πλήγμα στην πρόταση. Και σε ό,τι αφορά στους ανεξάρτητους πολιτές ασφαλιών, ασφαλίσεων και την πρόταση να αφαιρεθούν οι προμήθειες. Για μας αυτό είναι ένα θέμα ορισμού του όρου independent, ανεξάρτητος. Τι σημαίνει αυτό. Για μας ένας διαμεσολαβητής, ένας μεσάζων, ο οποίος λαμβάνει προμήθεια, με σημεριζολογικούς όρους δεν εμπίπτει στον ορισμό του ανεξάρτητου. Είναι ένα σημεριζολογικό ζήτημα λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα των μεσαζόντων ασφαλίσεων, αυτό είναι ένα παράδειγμα των τομέα που υπάρχει τάση να αφαιρείται η εξουσία της Κομισιόν για να υιοθετεί κατεξουδότηση πράξης. Χωρίς να αναφέρω τα υπέρ και τα κατά, θα αναφέρω ένα οριζόντιο ζήτημα, ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουμε τροπολογία που προτείνει να αφαιρέσουμε την εξουσία της Κομισιόν Εθετή κατά εξουσιοδότης πράξης, το λογικό είναι ότι ταυτόχρονα θα, προταθεί, θα προταθούν όλες οι λεπτομέρειες που θα καλύπτονταν με τις κατά εξουσιοδότης πράξης σε επίπεδο ένα της πρότασης. Η Κομισιόν προτείνει κατά εξουσιοδότης πράξης επειδή χρειαζόμαστε λεπτομέρειες διατάξεις Επομένως, ορισμός ε, των σωστών επαγγελματικών προσόντων για τις δυσυνοριακές ε, δυνατότητες των αστυνομικών ασφαλίσεων είναι ένα παράδειγμα. Αν λοιπόν πάει στο επίπεδο 1 του κειμένου, χρειαζόμαστε λεπτομερείς διατάξεις για το ποια θα ήταν τα αποδεκτά προσόντα. Και υπάρχουν και οι έννοιες δέσμευσης και ομαδοποίηση θα ήταν επιθυμητό να διασφαλίσουμε στους κανόνες σε όλη την αγορά, να έχουμε παραλληλισμό με την πρόταση MIFID. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι προσθέζεται εδώ στο MIFID. Για να συνοψίσω. Λοιπόν, είναι μια πρόταση που έχει ως στόχο την προστασία του καταναλωτή. Δεν πιστεύουμε ότι επιβάλλει υπερβολικό άχθος ε, στις ΜΜΕ και η πλήρης κάλυψη των διάβλων πώληση για την ασφάλιση και πλήρη διαφάνεια για τις αμοιβέ χωρίς έτοιμα ε, από τον πελάτη είναι στοιχεία που θεωρεί η Κομισιόν στο επίκεντρο της πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιεκτική σας απάντηση για τα θέματα αυτά. Να δώσω τότε το λόγο στην κυρία Στάιλερ για να συνοψίσει και να σχολιάσει αυτά που υπόθηκαν και μετά να μας πει και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κοιόδες εισηγητές. Εγώ νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, θέλουμε να είναι βελτιωμένη η προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτό και συμφωνώ με αυτό που, είπαν, που είπε η Επιτροπή αλλά και άλλοι για την ευθυγράμμιση με την πρόταση MIFID. Μπορεί να υπάρχουν ε, σύνδεσμοι και σε σχέση με αυτό που ο κύριος Χάβερ για, την, ε, για τις συμβουλές. Δεν θέλουμε να υπάρχουν συμβουλές όταν δεν απευθύνονται στον πελάτη, στον καταναλωτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Καμιά φορά η καθοδήγηση, οι συμβουλές είναι απλώς επεξήγηση του προϊόντος και όχι πραγματική συμβουλή. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε όταν το συζητούμε αυτό ότι υπάρχει σαφήνεια. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι όταν εμείς προωθούμε τις δικές μας ιδέες για την προστασία των καταναλωτών, που φανταζόμαι ότι είναι τελείως διαφορετική από αυτά που προτείνει η Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ενθαρρύνουμε και δεν αποδυναμώνουμε ε, την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Έχουμε κάποια στοιχεία μπροστά μας εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να γίνει μία ακόμη συνάντηση των σκιωδών ε, πριν από την ψηφοφορία που θα γίνει στις 25 Απριλίου. Είναι δυνατόν την επόμενη εβδομάδα να γίνει μία συνάντηση σκιωδών εισηγητών στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλύτερο γιατί περισσότεροι θα είμαστε εκεί. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, προτείνω 23 Απριλίου. 23 Απριλίου κάτι που μας δίνει δύο μέρες μέχρι την ψηφοφορία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τις συμβιβαστικέ πριν από τις 23, αλλά αν δεν υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε στο Στρασβούργο, τουλάχιστον Μία τελευταία συνάντηση σκιωδών θα ήταν πολύ χρήσιμη πριν από την ψηφοφορία με όλους όσους ε, ε, συμμετέχουν ε, στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθειά σας. Δεν είναι εύκολο τομέας από απόψε ως περίπλοκων στοιχείων. Και επίσης ε, υπάρχει και παραπομπή σε άλλες οδηγίες. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα συνάδουν με αυτά που έχουμε ε, γράψει. Ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες των συναδέλφων. αν υπάρχουν ε, στοιχεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε ώστε να ε, είναι σαφέστερη η διατύπωση. ευχαριστώ να συμπεριλάβω. Έχουμε ήδη κάποιες ε, τροπολογίες συμβιβαστικέ, 16 τον αριθμό, που ελπίζω να μας βοηθήσουν πολύ μέχρι την ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όντω ε, το χρονοδιάγραμμα το θέτουμε για να έχουμε μια συζήτηση εκ των προτέρων για τι συμβιβαστικέ τροπολογίε όταν ο κόσμο θα έχει τη δυνατότητα να τι διαβάσει. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο να τι έχουμε το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Κάρας που είναι βέβαια ο βασικό ε, ε, φαντάζομαι ότι θα το προωθήσει. Να περάσουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα το πρωί για τα, για τα έγγραφα με βασικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα. Ο κύριος Κοφεράτη θα εκπροσωπήσει τον κύριο Παντσέρη σήμερα και η κυρία Κόλιν Λάγκεν την κυρία Πιετικάινεν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, θα μιλήσει για τον κύριο Μπουζόη. Όχι γνέφει ο κύριος Χατζημαρκάκης, είναι εδώ και εκπρόσωπο τη ΓΚΟΕ. Θα ε, ζητήσω και την άποψη των σκιωδών εισηγητών. Πρώτο όμω, ο κύριος Κοφεράτη να μας παρουσιάσει το πακέτο συμβαστικών τροπολογιών του κυρίου Παντσέρη. Μετά ο κύριος Λίντερ Επίση θα πάρει το λόγο και θα ολοκληρώσουμε στις 12.30. Ε, Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο, εκ μέρους του κύριου Παλτσέρη αποσιάζει επειδή έχει ορισμένα καθήκοντα ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας με τις χώρες του Μαγκρέπο. Αντώνιο. Με παρακάλεσε να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει μέχρι εδώ, κάτι που το κάνω με ικανοποίηση. Από την τελευταία συνεδρίαση που έλαβε χώρα, με τους σκιώδεις εισηγητές πρόκειψαν κάποιες ε, παρατηρήσεις για ορισμένες από τις συμβιβαστικές λύσεις που είχαν ε, προσδιοριστεί προηγουμένως. Ο Αντώνιο συνέταξε εκ νέου τους ε, συμβιβασμούς λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συναδέλφων και τώρα θα σας συνοψίσω τις ε, τελευταίες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά το συνδεσμό G. Απλουστεύτηκε η διατύπωση σε σχέση με το πρόσθετο κόστος που δεν παρουσιάζεται στο εσωτερικό kit. Για το Συνδεσμό EI επαναβεβαιώθηκε η πρόταση που προβλέπει η Κομισιόν να επικυρώσει τεχνικά πρότυπα που έχουν εκπονήσει κύριες εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και αυτά να επαληθευτούν ε, με την Συμβουλή των Καταναλωτών δηλαδή πριν υιοθετηθούν. Σε ό,τι αφορά το σύστημα ταξινόμησης του κινδύνου, η πρόταση είναι αυτή ενός ε, γραφικού μοντέλου έγχρωμου για να μπορεί να συγκριθεί με αυτό που χρησιμοποιείται για στον τομέα της ενέργειας. Αυτό το μοντέλο που ε, είναι αντικείμενο έμπνευση από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην Πορτογαλία, που χρησιμοποιείται και καιρό στην Πορτογαλία, αποτελεί ένα καλό συμβιβασμό, σύμφωνα με τον συγκητή μεταξύ αυτού του πολύ απλού, με το φωτεινό συμβατοδότη και αυτού του ιδιαίτερα πολύπλοκου που χρησιμοποιείται στην ε, οδηγία για το συμβασμό G. Εδώ έχουμε το συμβασμό συνοχής μεταξύ της ε, ε, ενημέρωσης που έχουμε στο KIT και των εγγράφων που έχουμε στο φυλάδιο για το συμβασμό ο ομικρών, σε σχέση με τον μηχανισμό Ελεκτική επίλυση διαφορών, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε αυτούς, ε, αυτά πιο λεπτομερώς ε, στο διατακτικό θα συμπεριληφθούν όλες οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν από τον κύριο Παντσέρη και, και γίνεται και μία αναφορά στην εφιστάμενη ε, και ζήτησε να γίνεται μάλλον μια αναφορά και στην ειστάμενη οδηγία είναι υπάρχει μια νέα παράγραφος για τα προκαθισμένα κατόφλια προκειμένου να αποφευθούν ενδεχόμενες καταχρήσεις ε, του μηχανισμού προσφυγής. Η συνάντηση που είχε προβλεφθεί για χθε, όπως ε, ξέρετε, ακυρώθηκε επειδή αναχώρησε ο συγχυτής. Όμως, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει τους και όδης αν το θεωρούν σκόπιμο να παρουσιάσουν εδώ τις ε, παρατηρήσεις τους. Εγώ δεν τις καταγράψω προσωπικά και κατόπιν θα τις διαβάσω τον κύριο Παντσέρη. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι σύμφωνα και με τη γραμματεία της Επιτροπής, ήδη έχει προβλεφθεί η οργάνωση μιας τελευταίας συνεδρίασης πριν από την ε, ψηφοφορία της 25ης Απριλίου Επομένως, θα μπορούσε εκείνη να αποτελέσει την ευκαιρία οι παρατηρήσεις ή τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών που τους ευχαριστώ του νέου να αναφερθούν ξανά. Ευχαριστώ πολύ που μας αναφέρετε τη σκέψη του κ. Παντσέρη, η κ. Κονιλάντη. Καταρχάς, εξ ονόματος της κυρίας είναι θα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία και τους συμβιβασμούς που παρουσίασε. Η πρόταση είναι απαραίτητη για την προστασία των καταναλωτών στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αυτό επίσης συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες και τους προτινόμενους συμβιβασμούς, Πιστεύω ότι σε πολλούς τομείς μπορούμε να συμφωνήσουμε, υπάρχουν όμως ορισμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να διευκρινιστούν. Η έννοια του κινδύνου και η παρουσίαση του προφίλ κινδύνου είναι κάτι που αποτελεί πρόκληση. Δεν είμαστε απολύτω πεπισμένοι με το πώ προτείνει η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Έπειτα, οι δείκτε κινδύνου και αξιολογήσει κινδύνου από τι προηγούμενε επιδόσει ίσω δεν είναι οι καλύτερε σε διότι σε πολλές περιπτώσεις είναι παραπλανητικές. Πολλά αποδεικτικά στοιχεία μας δείχνουν ότι η παλαιότερη απόδοση δεν είναι χρήσιμη ένδειξη για το πώς ένα προϊόν θα αποδώσει στο μέλλον. Επίσης, όσον αφορά το PRIPS, ο κίνδυνος που συνδέεται με οποιοδήποτε προϊόν είναι έχει μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με το προϊόν και αυτό πρέπει κάπως να φανεί και στο κείμενο. Μία βελτίωση ενδεχομένως είναι να συμπεριληφθούν και τα διάφορα σενάρια κινδύνου όπως προτείνει ο εισηγητής. Ωστόσο δεν θα ήθελα να περιοριστώ σε απλά απαρίθμηση πιθανότητων, αλλά πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα τραπεζικά λιανικά προϊόντα, προσέχοντας όμως να μην είναι παραπλανητικό και πιστεύω πως ε, τα, η ταξινόμηση αναχρώμα ίσως είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα, ε, κάτι που συνδέεται με διαφορετικά είδη κινδύνου λόγω της ε, περίπλοκης ε, τους. Πρέπει να γίνει σαφές ποιο είναι δηλαδή το κόστος που συνδέεται με κάποιο πώς, ε, το κόστος που συνδέεται με κάποιο ταμείο. Επίσης, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε τη πληροφορία αυτή ξεχωριστά σε ένα άλλο σημείο. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της νομοθεσία, προτείνουμε να μην καλύπτει μόνο αυτά τα προϊόντα, αλλά όλα εν γέννη τα προϊόντα λιανικής. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στα επενδυτικά προϊόντα και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά ομόλογα θα συμπεριλαμβάνονται και να αποφευθούν οι παραπλανητικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Με τα κρατικά ομόλογα, από τα κρατικά ομόλογα προκύπτουν πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα με την διάδρασή τους με άλλα ομόλογα. πολλοί επενδυτές που επενδύουν σε προϊόντα λιανικής έχουν έλλειψη πληροφοριών. Πληροφορίες που έχουν δεν ε, επαρκούν. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη πληροφόρηση των πιθανών επενδυτών. Και να έχουν επιλογή από διάφορα ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χέντελ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Παντσέρη, ο συνάδελφος τον οποίο αντικαθιστώ. Είναι μια πολύ καλή βάση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, πιστεύω. Υπάρχουν ορισμένοι, ορισμένα σημεία τα οποία για εμάς είναι δύσκολα και θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε μια συνετή λύση. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουμε όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Εμείς θεωρούμε πολύ Θεωρούμε ότι αυτή η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα και να συγκρίνουν τα διαφορετικά προϊόντα. Επίσης, το ζήτημα της ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Χρειάζονται αποδείξει. Επίση, τι γίνεται με τι ε, κυρώσει σε περίπτωση που κάποιο δεν συμμορφώνεται με την οδηγία. και η σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών επίσης, ε, με τρόπο σαφή και εφεδιάκριτο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο έχει πολύ μεγάλο κόστος, όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν διάφανη και καλύτερη ενημέρωση και ίσως αυτό θα γίνει εάν επικεντρώνεται η εκάστοτε ενημέρωση σε συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν και να μην είναι τόσο γενική. Τώρα όσον αφορά τους δείκτε κινδύνου, το θεωρούμε μια πολύ καλή ε, επιλογή, μια πολύ καλή δυνατότητα να υπάρχουν αυτοί οι δείκτες έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να πληροφορείται για τους κινδύνους. Φυσικά αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ε, απλούστερη και κατανοητή. και οι κίνδυνοι πιστεύουμε πως πρέπει να είναι έτσι παρουσιασμένοι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τους συγκρίνει πολύ εύκολα και να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαφάνεια. Ο καταναλωτής είναι πλέον σε θέση να απαιτεί, να μάθει και να γνωρίζει πού επενδύει. Ευχαριστώ. Ναι, συμμερίζομαι τις απόψεις σας. Ωστόσο ξέρω ότι στο συμβαστικό άρθρο 6 εσείς μιλάτε για έναν σύντομο και περιεκτικό τρόπο που δεν θα ξεπερνά τις τρεις σελίδες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αντιφατικό ως έχει. Δηλαδή τις σελίδες α4. Δεν είναι τόσο σύντομο αυτό. θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο για να διαβάσουμε όλες τις ενημερω... ενημερωτικές σημειώσεις σας, αν είναι τόσο πολλές. Όμως, γνωρίζουμε για τους ε, περιορισμούς και το πόσο περίπλοκη είναι η πληροφόρηση των ε, καταναλωτών. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό σε αυτήν την Επιτροπή στο παρελθόν και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε. Επίσης, αυτές οι συνοπτικές πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως ορισμένα επισημασμένα σημεία. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω τι θα είχε να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας. Ε, εάν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος άλλος θα ζητήσω να πάρει το λόγο η Επιτροπή και να μας πει πώς βλέπει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους ε, εισηγητές και τους κοιόδες εισηγητές. Ευχαριστούμε πολύ που η Επιτροπή στηρίζει την πρότασή μας τόσο πολύ. Και είδαμε τις τροπολογίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύουμε πως πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. φυσικά είναι και πολύ σημαντικό θέμα. Όταν ορίζουμε το πεδίο εφαρμογή στα, στη δέσμη προϊόντων. Το κάναμε αυτό διότι αυτά τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και δεν μπορούν να τα καταλάβουν εύκολα οι καταναλωτές. Κατανοούμε τη συζήτηση για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή και είναι εύλογο το έτοιμά σας. Όμως εάν διευρυνθούμε πάρα πολύ τότε θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα είναι δύσκολο και δεν θα είναι πλέον απλό, διότι η δομή θα πρέπει να, ε, να τεντώσει για να πάρει όλους τους ορισμούς. Αυτό θα κάνει πολύ περίπλοκο και πολύ πιο δυσνόητο το κείμενο. Επίσης, μια άλλη βασική ιδέα που αναφέρεται το πόσο σύντομο πρέπει να είναι το κείμενο, το πόσο μικρό. Έχουμε εμπειρία από το παρελθόν για το πώς το κάνουμε αυτό. Προτού όμως ορίσουμε επακριβώς το περιεχόμενο, πρέπει να γίνουν εκτενείς έρευνες πάνω σε καταναλωτές και μελέτες τώρα όσον αφορά το μέγεθος, την έκταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως αυτά πρέπει να γίνουν σε πράξη επίπεδου 2, διότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν με τόση λεπτομέρεια σε μια οδηγία. Τώρα, κάποιες άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται στις τροπολογίες, να πω ότι εμείς δεν διαφωνούμε αλλά το θεωρούμε πως είναι καλύτερο να, θεωρούμε πως είναι καλύτερο να μπουν σε πράξεις επίπεδου 2 λόγω του λεπτομερούς χαρακτήρα, διότι πιστεύουμε πως στο κείμενο αυτό στην οδηγία θα παρεμποδίσουν την σωστή λειτουργία της και εφαρμογή της. Γι' αυτό προτείνουμε λοιπόν να πάει από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 2, όπως προβλέπετε εξάλλου. Επίσης, Φυσικά και μας ενδιαφέρει ο ρόλος του, του μεσάζοντα και ο ρόλος του παρόχου. Ο πάροχος, για παράδειγμα, διαχειρίζεται ένα ταμείο και σε συνεργασία με έναν μεσάζοντα. Ποιος όμως έχει την ευθύνη. Έχουμε κάνει πολλές σκέψεις γι' αυτό. Και θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερωθεί και να ενημερωθεί από ένα απλό κείμενο και αυτό φυσικά εμπεριέχει ευθύνη για, τον, εκείνον που παράγει ένα προϊόν και το θέτει στην αγορά αλλά και για εκείνον που το αγοράζει όμως. Και είναι πολύ σημαντικό ο καταναλωτής να μπορεί να απευθύνεται είτε στον μεσάζοντα είτε στον παραγωγό με απλό τρόπο. Τώρα όσον αφορά τα συστήματα προειδοποίησης και αυτό που είπατε εσείς για το φανάρι με τα τρία χρώματα, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, ναι, είναι, κάνουμε λίγο μαγικά έτσι όπως το λέτε. Έχουμε πολύ δύσκολα προϊόντα τα οποία προσπαθούμε να συνοψίσουμε και να τα περιγράψουμε με πολύ απλό τρόπο. Δεν είναι αδύνατον, είναι όμως πολύ δύσκολο. Και αυτά τα συστήματα προειδοποίησης θα μας βοηθήσουν. Όντως, πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην υπεραπλουστεύσουμε κάτι που είναι από τη φύση του αρκετά περίπλοκο. Γι' αυτό θα προτιμούσαμε αυτές οι λεπτομέρειες να επεξηγούνται μαζί να, ε, να επεξηγούνται αφού έχουν γίνει όλα τα τεστ και όλες οι έρευνες πάνω σε καταναλωτές και σε συνεργασία με την ΕΣΠΑ. Δεν θα προτιμούσαμε να έχουμε εδώ τόσες πολλές λεπτομέρειες, θα προτιμούσαμε αντίθετα να έχουμε την ελευθερία να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Βέβαια πάντα σε συμφωνία με, τις, ε, με τη Γενική Αρχή που θα διέπει το κείμενο. Αυτά νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ περιεκτικός και συμφωνούμε και με αυτό που είπατε σε σχέση με τις δοκιμές ε, των καταναλωτών ε, για να είμαστε βέβαιοι ότι περνάει με αποτελεσματικό τρόπο το μήνυμα στους καταναλωτές γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Κύριε Κοφεράτη, μήπως θέλετε να σχολιάσετε τίποτα, να μας πείτε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Όχι, μόνο μια γρήγορη σκέψη. Η χρόνη είναι αυτή που είχα πει προηγουμένως. Θα έχουμε αυτή την μετέπειτα συνεδρίαση με τους κοιόδης, εισηγητές, πριν από την ψηφοφορία που προτείνεται για τις 25. Η μόνη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι εξή. Φυσικά θα διαβιβάσω στον κύριο Παντσέρη τις παρατηρήσεις σας, ακριβώς έτσι όπως τις διατυπώσατε. Το πεδίο εφαρμογή είναι ένα θέμα όχι μόνο κεντρική σημασία, αλλά και λεπτό. Όμως ήθελα να σημειώσω ότι αν είναι αλήθεια ότι αν ε, μια υπερβολή επέκταση μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη διαχείριση, είναι και αλήθεια ότι μια λογική επέκταση του πεδίου εφαρμογή βάζει τον καταναλωτή σε θέση να έχει περισσότερα προϊόντα να συγκρίνει και όταν ένα άτομο μπορεί να αξιολογήσει τις διαφορές ε, και να κάνει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων, ε, γνωρίζει πολύ καλύτερα τελικά ποια επιλογή θα κάνει. Είναι πολύ πιο συνειδητή η επιλογή του. Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή. Όπως είπαν και αρκετοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ και πάλι και θα παραπέμψω τις παρατηρήσεις σας στον συγητή. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αντικαταστήσατε τόσο αποτελεσματικά τον κύριο Παν, ε, Παντσέρη. Οπότε, συνεχίζουμε. Θα εγκρίνουμε την ογνωμοδότησή μας με όλους τους συμβασμούς στις 25 Απριλίου. Μετά η αντίστοιχη ημερομηνία στην ΕΚΟΝ είναι το Μάιο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά μπορούμε κάτι να κάνουμε στον διάμεσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε έτσι τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήταν εδώ να μας εξηγήσει ε, περισσότερα και μας έδειξε και την εμπειρογνωμοσύνη της. Η επόμενη μας συνεδρίαση είναι στις 24 και 25 Απριλίου, τέσσερις συνεδρίες ε, 9 το πρωί και τελειώνουμε 6.30 την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους αλλά και όσους μας ακούν στο διαδίκτυο. Ελπίζουμε και στο μέλλον να μας ξαναπαρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πέρα τη συνεδρίαση.